Buenos días. Καλημέρα σας. Καθίστε παρακαλώ. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Ε, continuamos con el orden del día. Λοιπόν, άρχεται η συνεδρίαση. Σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Οι συντονιστές χρειάστηκε να καθυστερήσουν λίγο. Πρώτο θέμα, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Σας παρακαλώ λίγη ησυχία. σας ενημερώνω ότι τα σημεία 4 και 6 εκθέσεις Αρσένη και Τωμά θα αναβληθούν και υπάρχει πρόταση και το 5 η συμφωνία με το Μπάτι να αναβληθεί σε συνεδρίαση των ε, συντονιστών η πλειονότητα όχι ομόφωνα σε συνεδρίαση των συντονιστών σας προτείνουν να αναβληθεί μέχρι τις 17 από ό,τι με ενημέρωσαν και να ζητήσουμε μια έκθεση που ούτως ή άλλως θα πρέπει να έχει ληφθεί πριν τις 17 και είτε έχει ληφθεί ή όχι θα ψηφιστεί αυτή η έκθεση στις 17. Αυτή είναι η πρόταση που ε, μου έγινε. Δεν ξέρω αν έτσι ακριβώς ε, έχουν τα πράγματα αν έχει κάποιος να πει κάτι. Προτείνεται λοιπόν να αναβληθεί με αυτές τις προϋποθέσεις αυτό το θέμα. Η κυρία Πατράου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Απλώς να επιβεβαιώσω, επειδή όλοι, ε, επειδή εγώ μάλλον είμαι κατά της αναβολής όπως όλοι το ξέρουν, στην συνεδρίαση που οργανώσαμε για να συμφωνήσουμε Είπαμε να πάμε στις 17 του Οκτώβρη να αποσταλεί το νομοθετικό έγγραφο, αλλά σε κάθε περίπτωση είτε φτάσει το έγγραφο γέρος είτε όχι, η ψηφοφορία θα γίνει. Δεν θα υπάρξει πλέον, επιπλέον αναβολή. Αυτή ήταν η συμφωνία μας. Και βεβαίως θα ζητήσουμε την νομική γνωμοδότηση και βάσει των πληροφοριών που έχουμε ως τώρα, θα φτάσει το έγγραφο στην ώρα του, αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που πάμε στην συνάντηση εκείνη, φτάσει δεν φτάσει, είτε υπάρξει συμφωνία από την νομική υπηρεσία είτε όχι, η ψηφοφορία θα γίνει στα 17. Έχουμε μόλι δύο εβδομάδε. Αυτή είναι η μόνη παραχώρηση που μπορώ να κάνω. Καμιά άλλη. Έτσι θα το κάνουμε, οπότε τροποποιείται η μερίσια διάταξη. Οπότε σήμερα δεν θα έχουμε ψηφοφορίες. Σημείο 3. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Δεν υπάρχουν. 4, 5 και 6 αναβλήθηκαν. Περνάμε λοιπόν. Δεν θα γίνουν ψηφοφορίες και περνάμε στο 7. Απόφαση του Συμβουλίου για πρωτόκολλο για να καθορίσουμε τους όρους αλληλείας και την οικονομική αντιστάθμιση για τη συμφωνία αλληλείας μεταξύ της Ένωσης και της ακτής τους 18 Ιουνίου κάναμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και σήμερα θα ακούσουμε τον κύριο Κωτινί το σχέδιο σύστασης που έχει υποβάλει. Παρακαλώ. Ο κύριος Κωτινί. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ό,τι αφορά τη συμφωνία αλλία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και έκτη του δεν βλέπω ιδιαίτερε δυσκολίε, Το έχω να κάνω ιδιαίτερε παρατηρήσει. Πρόκειται για μια εταιρική σχέση που έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70. Οι τελευταίε διαπραγματεύσει έγιναν σε κλίμα φιλικό και με μεγάλη ταχύτητα. Ε, το πρωτόκολλο θα ισχύσει προσωρινά από την 1η Ιουλίου του 2013 και θα ισχύει ω τι 30 Ιουνίου του 2018. Υπάρχουν αλλιευτικέ δυνατότητε για το γαλλικό και ισπανικό στόλο, πιο συγκεκριμένα για 28 ε, ε, και για παραγαδιάρικα επιφανία. Σε ε, οικονομικό επίπεδο η αντιπαροχή φτάνει τα 620.000 ευρώ τον χρόνο, 257.000 για την πρόσβαση ε, σε, στα ύδατα της χώρας. η τόνοι φτάνουν περίπου τους 600.000 τόνους ετησίως και σε σχέση με το προηγούμενο πρωτόκολλο βλέπουμε να υπάρχει αύξηση στην οικονομική ε, αντιπαροχή και μείωση του συνόλου των τόνων. Αυτό για να προστατευτούν τα, οι ελευτικοί πόροι. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι οι ελευτικές δυνατότητες σήμερα είναι πλέον απορκετές, περισσότερο απορκετές. Σε κοινωνικό επίπεδο είναι ενδιαφέρον το πρωτόκολλο και για τις δύο πλευρές, διότι τα σκάφη ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολούν πλέον 20% περισσότερο ψαράδες από την Αφρική και βεβαίω ε, αυτό είναι καλό και για του πλειοκτήτε τη ε, Ευρώπη. Είναι σημαντικό το πρωτόκολλο για την ανεξαρτησία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που όπω θυμάμαι είναι ο πρώτο εισαγωγέα διεθνώ ελευμάτων Ελπίζουμε λοιπόν οι Περιφερειακέ Επιτροπέ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσουν για του ελευτικού πόρου και τι εντηρήσει του. Να θυμίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα επιθυμούσαν να ενισχύσει του ελέγχου για την ε, χρήση κάποιων εργαλείων στην ε, ακτή του ελεφαντοστού και ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει επίση να παρακολουθήσει την υλοποίηση τη συμφωνία και καλό θα είναι να γνωρίζει πώ εξελίσσονται τα πράγματα στην πράξη. Να προσθέσω ότι επιτροπέ ανάπτυξη και προπολογισμών τάθηκαν υπέρ του πρωτοκόλλου αυτού και δεν έχω ιδιαίτερε παρατηρήσει για την κύρωση του πρωτοκόλλου, ούτε αντιρρήσει από το Κοινοβούλιο. Σα προσκαλώ λοιπόν να το εγκρίνουμε. Ευχαριστώ. Muchas gracias, eh, señora Ευχαριστώ κυρία Μάσινα. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Είναι συνέχιση ενός ε, πρωτοκόλου που υπάρχει από το 1990 και για τις δύο πλευρές ε, είναι πολύ ισορροπημένο. Πρέπει να πληρώσουμε λίγο περισσότερο, μπορούμε γι' αυτό βέβαια να αλλιεύουμε λίγο λιγότερο, αλλά σέβεται τις αρχές της αναπτυξιακής μας πολιτικής που λέει ότι οι εταίροι μας πρέπει να έχουν δυνατότητα να αναπτύξουν το δικό τους τομέα και εμείς βέβαια να έχουμε κάποια δικαιώματα για τους αλληλείς μας από την Ισπανία και τη Γαλλία. Πρόκειται κυρίως για ε, αλληλεία τόνου που μας ενδιαφέρει πολύ. Είναι πολύ ισορροπημένο, όπως είπε ή μάλλον όπως έγραψε, δεν είπε ο εισηγητής, στην ε, ακτή ελεφαντοστού υπάρχουν ε, ταραχές αυτή τη στιγμή και κάποια σταθερότητα σε αυτό το τομέα θα μπορούσε να βοηθήσει τη χώρα οικονομικά να σταθεί στα πόδια της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος. Δεν θέλει άλλο το λόγο. Ποιο θα μιλήσει. Α, όχι, κυρία Πατράω. Πολύ σύντομα, απλώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου που σήμερα συζητούμε τρεις ε, συμφωνίες. Κάτι που στην πραγματικότητα ουσιαστικά εδρεώνει την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διαφορετικές περιοχές ε, της θάλασσας του κόσμου, των θαλασσών του κόσμου. Ε, και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εκεί που δεν θα βρεθούμε εμεί, άλλοι θα καλύπταν τη θέση μα. Γι' αυτό πρέπει να αναλάβουμε τι ευθύνε μα και τι ε, υποσχέσει που έχουμε δώσει να τι εκπληρώσουμε για την κοινωνική εξέλιξη των χωρών με τι οποίε συνάπτουμε συμφωνίε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με την ακτή του Ελεφαντοστού είναι σαφέ ότι όλε οι, οι απαραίτητε εγγύσει έχουν δοθεί μέσω του πρωτοκόλλου και μπορούμε να πούμε και σε συνέχεια των όσων επιβεβαίωσε και η ακτή του ελεφαντοστού ότι εκφράστηκαν κάποιες απαιτήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτές πρέπει όλο και περισσότερο να συμπεριλαμβάνονται στις νέες μορφές συμφωνίας. Προφανώς υπάρχει κάποια μείωση στις αλληλευτικές δυνατότητες και μια αύξηση του οικονομικού αντιτίμου της αντιπαροχής, όμως δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά, οπότε δεν νομίζω να αποτελεί πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πατράου. Η Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Δεν έχω να προσθέσω και πολλά. Συμφωνώ πλήρω με την εισηγήτρια. Μπορώ επίση να σα διαβεβαιώσω ότι συνεργαζόμαστε στενά με την κυβέρνηση της ακτή Ελεφαντοστού έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε όλοι να συνεργαστούμε, να αναπτυχθεί ο τομέας τους, να παράσχουμε τεχνική βοήθεια και τεχνογνωσία ε, πέρα από την οικονομική βοήθεια. Πρόκειται λοιπόν για μια συμφωνία στο πλαίσιο της οποίας θα έχουμε μια στενή συνεργασία και θα είναι αμοιβαία ε, επωφελής και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ακτή Λεφαντοστού. Ευχαριστώ. Οπότε Έληξε συζήτηση, προθεσμία υποβολής τροπολογιών 8 Οκτωβρίου 12 ώρα το μεσημέρι και η ψηφοφορία θα γίνει τον Νοέμβριο. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, το 8, πρωτόκολλο Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου για τον καθορισμό των αλληλευτικών δυνατοτήτων. Στις 18 και 19 Ιουλίου υπεγράφει στο Ραμπάτ ε, το πρωτόκολλο αυτό, η Κομισιόν μας υποβάλλει την πρόταση και πρώτα θα ακούσουμε την πρόταση της Επιτροπής και κατόπιν θα ακούσουμε την κυρία Φράγα, την εισηγήτρια. Ε, ο κύριος ε, Ντεμπιπέρ, από πλευρά της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ας το θέσω έτσι, ανταποκριθήκαμε στο αίτημα του Κοινοβουλίου της Επιτροπής Αλίας. Όταν είχε συνδεθεί το προηγούμενο πρωτόκολλο, είχατε απορρίψει την πρόταση της Επιτροπής, γιατί δεν θεωρήθηκε ικανοποιητική από πλευράς σχέσεις κόστους-οφέλους. Και τότε λοιπόν μας είχατε ζητήσει να επανέλθουμε στις διαπραγματεύσεις και να διαπραγματευτούμε ένα καινούριο πρωτόκολλο, το οποίο θα διόρθωνε τα προβλήματα της α, χαμηλής χρήσης, της και μας ζητήσατε το νέο πρωτόκολλο στο οποίο θα καταλήγαμε να είναι επωφελές και από οικονομική και από ε, περιβαλλοντική πλευρά και για, τα δύο μέρη. Και ταυτόχρονα να εγγυηθούμε ότι το, η αλληλεία θα αφορά μόνο στο πλεόνασμα το οποίο πλεόνασμα θα πρέπει να παρακολουθείτε στενά και αποτελεσματικά. Επίσης ζητήσατε να υπάρξει μια ρήτρα ανθρωπινών δικαιωμάτων. Προς όφελος του πληθυσμού, του, του λαού του Μαρόκου. Η εντολή που μας έδωσε το Συμβούλιο ήταν πάνω κάτω ίδια. Μας έθεσε πάνω κάτω τους ίδιους όρους. Και ε, από αυτή τη βάση διαπραγματευτήκαμε με την κυβέρνηση του Μαρόκου. Πιο ε, ικανοποιητική λοιπόν σχέση κόστους κόστους-οφέλους, μεγαλύτερη ε, λήψη υπόψη της, των επιστημονικών δεδομένων για το περιβάλλον. Ταυτόχρονα βέβαια η αναθεώρηση της πολιτικής που διεξήχθη στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε στο να υπάρξουν και άλλες ε, προϋποθέσεις που έχουν σχέση με την αναθεώρηση της πολιτικής ε, εξωτερικής δράσης, όπως ε, για παράδειγμα η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ρεσιμότητα βάση αυτής. Σας παρουσιάζουμε λοιπόν την πρότασή μας, την οποία πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται σε αυτό που μας ζητήσατε. Δεν σας παρουσιάσω όλε τι λεπτομέρειε, μόνο κάποια σημαντικά στοιχεία τη συμφωνία. Οικονομική αποτελεσματικότητα. Πιστεύω ότι αυτό το πετύχαμε αυξάνοντας τι δυνατότητε αλλίευση κατά 33% περίπου. Και το σημαντικότερο στοιχείο νομίζω είναι η βιομηχανική πελαγική αλληλεία που τώρα θα ανέρχεται στους 80.000 τόνους. Ε, επίσης δόθηκε δυνατότητα για περισσότερα ε, αλλιευτικά παραγαδιάρικα βυθού στο βορρά, ανάμεσα στα άλλα. Και πάλι όσον αφορά την οικονομική αποτελεσματικότητα, καταφέραμε να μειώσουμε την οικονομική βοήθεια για την πρόσβαση κατά 10% περίπου. Δηλαδή φτάσαμε στο, από τα 22,6 στα, ε, στα 16 εκατομμύρια. Και μειώθηκε η επιβάρυνση του κοινοτικού προπολογισμού κατά 17%. Συνολικά η οικονομική βοήθεια, η επιβάρυνση μάλλον για την ευρωπαϊκή οικονομία αυξάνεται, αλλά αυτό οφείλεται στην αύξηση των εισφορών από τους εφοπλιστές, από τους ε, αλής. Άρα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, καταφέρνουμε να έχουμε περισσότερες δυνατότητες με λιγότερο κόστος. Ένα μέρος του κόστους το επομίζονται οι εφοπλιστές. Επίσης βελτιώθηκαν οι τεχνικές προϋποθέσεις. Αν θυμάστε ε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα με την προηγούμενη συμφωνία ήταν, ήταν το ότι ενώ έδινε ε, δυνατότητες αλίες, οι τεχνικές προδιαγραφές δυσχέρεναν την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων. Βελτιώσαμε λοιπόν αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές και ε, κάναμε μια πολύ λεπτομεριακή ανάλυση σε συνεργασία με τους συναδέλφους από το Μαρόκο. Να σας αναφέρω ένα στοιχεία. Είναι η μείωση του αριθμού των ναυτών, ε, ε, επέκταση ε, δυνατοτήτων αλίας στο βορρά. Ήταν αρκετά διαλλακτικοί οι συνομιλητές μας από το Μαρόκο και θα μπορούσαμε να τα βελτιώσουμε αυτά τα στοιχεία ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Όπως σας είπα επίσης έχει αυξηθεί ο αριθμός των ε, σκαφών βιομηχανικής πελαγικής αλίας που θα έχουν τη δυνατότητα να αλλιεύουν ταυτόχρονα. Αυτό είναι τεχνικό αλλά σημαντικό. Επίσης για τα αλλιευτικά με ψυχτικές εγκαταστάσεις αυξάνεται η περιοχή στην οποία μπορούν να αλλιεύουν. Και όσον αφορά τη ναι, είναι σημαντικό αυτά τα σταλιευτικά να βρίσκονται κοντά στην ακτή γιατί ε, ε, χρειάζεται να απορρίψουν την αλία τους, το αλίευμα ε, άμεσα για επεξεργασία στην ακτή. Επίσης πολλά κρατημέλη ζήτησαν να παρακολουθούμε πιο στενά την, ε, τις ποσότητες που αλλιεύονται. Τώρα έρχομαι στο ζήτημα του, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και του, ε, της παρακολούθησης αυτού του στοιχείου. Αναφέρονται πολλά τέτοια στοιχεία όπως η βιώσιμη διαχείριση της αλληλείας στην συμφωνία, η ε, συνεργασία με το, με το Εθνικό ε, Ίδρυμα ε, Αλληλία στο Μαρόκο, το οποίο, με το οποίο συνεργαζόμαστε καλά και το οποίο έχει και καλό έργο. Οι εμπειρογνώμονές μας θεωρούν ότι λειτουργεί ε, σωστά αυτή η συνεργασία και θα τη συνεχίσουμε. Υπάρχει ένα στοιχείο καινούριο, η ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων. Αυτό θα αυξήσει την αξιοπιστία των στοιχείων. που είναι σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το Μαρόκο. Επίσης μας ικανοποιεί το γεγονό ότι αυτή η συμφωνία ταιριάζει με την γενικότερη στρατηγική μας. Και άρα ε, δεν αναφέρεται μόνο σε αυτό που θα κάνουν τα ευρωπαϊκά σκάφη, αλλά γενικότερα τα σκάφη στην περιοχή. Ταιριάζει με τη στρατηγική μας για την περιοχή. Επίση, μα ικανοποιεί το γεγονό ότι το Μαρόκο αναλαμβάνεται και δεσμεύεται να ε, ε, ε, συνεργαστεί στην καταπολέμηση τη παράνομη αλεία. Επομένω, θεωρώ θετικό βήμα στην ενίσχυση τη συνεργασία με τον Μαρόκο αυτό το πρωτόκολλο. Τέταρτο σημείο. Ικανοποιητικό. Το ζήτημα του στόλου ένα από τα προβλήματα της προηγούμενης συμφωνίας, η συνεισφορά μάλλον των εφοπλιστών. Στην προηγούμενη συμφωνία ήταν πολύ μικρή. Και αυτό δεν έδινε κίνητρα για αξιοποίηση της συμφωνίας. Τώρα με τη νέα συμφωνία οι ε, εφοπλιστές, οι αλληλείς πραγματικά θα συνεισφέρουν σε όλους τους το σε όλα τα είδη. Για την αλία μικρής κλίμακας, αυτή η αύξηση της οικονομικής συνεισφοράς είναι μικρή, αυξάνεται αλλά λίγο, αλλά όσον αφορά τη βιομηχανική αλία, εκεί φροντίσαμε η αύξηση να αντιστοιχεί στις αυξημένες αλληλευτικές δυνατότητες που τους δίνουμε. Θα διαπιστώσετε λοιπόν ότι η αύξηση τη συνεισφορά για την βιομηχανική αλληλεία είναι πιο μεγάλη από εκείνη για την αλληλεία μικρή κλίμακα. Υπάρχει επίση και μια άλλη διαστρωμάτωση. Για τα, τα μικρότερα σκάφη ζητάμε μικρότερη ε, ε, συνεισφορά. Ενώ ας πούμε για τα, για τα σκάφη με παρασυρώμενα δίχτυα ζητάμε να ε, συνεισφέρουν περισσότερο. Τώρα, το ζήτημα της ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, και τονίζουμε τη σημασία του με το γεγονό ότι το έχουμε βάλει στο πρώτο άρθρο συνδέεται επίσης με την Συμφωνία Σύνδεσης του 1996, η οποία αναφέρεται στις, ε, στις ανθρώπινα δικαιώματα και στις αρχές της δημοκρατίας. Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των αρχών προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής του πρωτοκόλλου με έναν μηχανισμό ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 8 του πρωτοκόλλου. Εκεί προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής του με πρωτοβουλία ε, ή του του ενός ή του του άλλου μέρους. Με άλλα λόγια δεν μας δεσμεύει αυτό το πρωτόκολλο, δεν μας εγκλωβίζει σε μια κατάσταση. Νομίζω ότι αυτό το επιθυμούσε και το Κοινοβούλιο. Επίσης κάτι άλλο που μας είχατε ζητήσει ήταν σεβασμός της διεθνούς νομιμότητας και να βεβαιωθούμε ότι ο τοπικός πληθυσμός υποφελείται και ότι θα υπάρχει λογοδοσία, θα υπάρχει, υπάρχουν εκθέσεις που θα δείχνουν πού δαπανώνται τα χρήματα. Αυτό προβλέπεται και θα υπάρχει μια ετήσια αξιολόγηση και μια μεικτή επιτροπή. Θα έχουμε ε, εκθέσεις για όλες τους τομείς της αλίας που θα καταγράφουν επίσης και τα κοινωνικά ε, αποτελέσματα στην, για παράδειγμα, απασχόληση, Επίσης προβλέπεται μια τελική έκθεση αλλά νομίζω πιο σημαντικό είναι ότι θα τα έχουμε αυτά τα στοιχεία σταδιακά. Δεν θα πρόκειται να περιμένουμε να λάβουμε μια έκθεση στο τέλος όλης αυτής, όλου αυτού του εγχειρήματο. Αντιθέτως, θα έχουμε τα στοιχεία αυτά ε, καθώς ε, προχωράει η υλοποίηση του πρωτοκόλλου. Κάποια άλλα στοιχεία είναι ότι ε, ε, αυτή η Αυτέ οι δραστηριότητες δημιουργούν ε, θέσεις εργασίας και δραστηριότητα και στην ακτή, δηλαδή δεν πρόκειται μόνο για αλληλεία. Αυτό, αυτή, αυτό το πρωτόκολλο θα ε, συμβάλλει, θα βοηθήσει και τον τοπικό πληθυσμό στις ακτές. Το ζήτημα της αρεσιμότητας της τομεακής ενίσχυσης και εδώ έχουμε ακολουθήσει την γενικότερη αναθεώρηση της πολιτικής μας για την αλληλεία. Έχει αποσυνδεθεί η τομιακή χρηματοδότηση. Ε, η τομιακή χρηματοδότηση γίνεται σταδιακά και υπό την αίρεση ότι έχουμε λάβει μια έκθεση η οποία θα αποδεικνύει ότι τα χρήματα αυτά θα δαπανηθούν όπως πρέπει ε, με τη γεωγραφική κατανομή που προβλέπετε και με την τομεακή κατανομή που προβλέπετε. Συνολικά λοιπόν το συμπέρασμά μου είναι ότι μετά από μια δύσκολη διαπραγμάτευση, μια επίπονη λεπτομοριακή ανάλυση όλων των στοιχείων, νομίζω ότι καταλήξαμε σε κάτι που ικανοποιεί και εμάς και τους ε, συνομιλητές μας στο Μαρόκο, γιατί που θα είναι επωφελές και για τις δύο πλευρές. Το νέο πρωτόκολλο είναι βελτιωμένο σε σχέση με το παλαιότερο, και νομίζω πετύχαμε αυτά που επιδιώκαμε. Κοιτώ λοιπόν αυτά που μας ζήτησε το Κοινοβούλιο και αυτά που μας ζήτησαν τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αποκριθήκαμε στις απαιτήσει σας. Και σας ζητώ λοιπόν να το εγκρίνετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Ντεπιπέρ η εισηγήτρια, κυρία Φράγα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Ντεπιπέρ. Να αρχίσω με αυτό που ε, ε, εκεί που κατέληξε. Μόλις ε, γύρισα από το Μαρόκο μετά από τη συνεδρίαση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις σχέσεις στον αλληλευτικό τομέα ή είχαν καλέσει σε μια συνεδρίαση στην Κάσα Μπλάνκα για να αποτιμήσουμε το πρωτόκολλο, αυτό το νέο πρωτόκολλο που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένη γιατί τόσο οι, μαροκινή Μαροκινοί στον τομέα αυτό και ο αλληλευτικός τομέας της Ένωσης ε, σε γενικές γραμμές είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό το πρωτόκολλο και όλοι το εκτιμούν θετικά. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ε, διαφοροποιήσεις, αποχρώσεις, αλλά γενικά πολύ θετική αποτίμηση. Και είχα τη δυνατότητα να μιλήσω και με τις αρχές που είναι υπεύθυνε για την αλληλεία στο Μαρόκο και αυτές είναι πολύ διατεθειμένε να συνεργαστούν μαζί μα, Ήδη συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μου υποσχέθηκαν ότι θα μα στείλουν στοιχεία που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην έκθεση και που θα ε, κάνουν ακόμη καλύτερο αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Και αυτά που είπε ο κύριος Ντεπίπερ. Δεύτερον, να υπενθυμίσουμε... όταν μιλάμε για Ηλία πάντα είναι καλό, ότι αυτό το νέο πρωτόκολλο εντάσσεται στο πλαίσιο των γενικότερων σχέσεων της Ένωσης με το Μαρόκο. Και από το 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χορηγήσει στο Μαρόκο ένα ε, καθεστώς. Πρώτη χώρα στην περίοδο της ε, Μεσογείου που θα μπορούσε να εντάξει το Μαρόκο σε μια εσωτερική αγορά εφόσον υπάρχει και η σύγκληση στο νομοθετικό και κανονιστικό τομέα. Υπάρχει λοιπόν ένα σύνολο σχέσεων με το Μαρόκο, το βασίλειο του Μαρόκου. Όπως θα θυμάστε, Ε, στην έκθεση Χάγκλουντ που ζήτησε να απορριφθεί στην Ολομέλη το 2011 η παράταση του πρωτοκόλου που ίσχυε προσωρινά για 8 μήνες και που τελικά απορρίφθηκε, όπως θα θυμάστε, στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου του 2011. Όπως θα θυμάστε λοιπόν σε αυτήν την έκθεση, είχα αναλύσει όλες τις επικρίσεις που είχαν διατυπωθεί και με ορισμένες φυσικά συμφωνούσα γιατί το προηγούμενο λοιπόν πρωτόκολλο είχε σοβαρά τεχνικά ελαττώματα. Θα θυμάστε ποιες ήταν οι τρεις βασικές πλευρές στις οποίες βασίζονταν οι επικρίσεις. Το οικονομικό θέμα, γιατί η ανάλυση κόστους ε, ε ήταν ε, ιδιαίτερα αρνητική. Το δεύτερο ήταν το περιβαλλοντικό, υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση των ε, αποθεμάτων, αλληλευτικών αποθεμάτων και το τρίτον ήταν ε, η πολιτική για τον κλάδο. Χαμηλή χρήση που είχε υπάρξει ε, από πλευράς των μαρακινών του προηγούμενου πρωτόκολλου. Ο εισηγητής είχε βασιστεί στο μόνο που είχαμε. Ήταν η έκθεση αποτίμησης εκ των υστέρων. Αυτή η περίφημη έκθεση που χρειάστηκε να μεταφραστεί κτλ και δύο χρόνια αργότερα η καινούρια ανάλυση και ιδιαίτερα σε σχέση με την έκθεση που είχαμε τότε όλα αυτά μας αποδεικνύουν ότι είχε εξεταστεί μόνο η περίοδος των ε, πρώτων 2,5 ετών εφαρμογής ε, της προηγούμενης συμφωνίας. Όχι λοιπόν όλη της περίοδου. Δεύτερον, με βάση τα επιστημονικά πορίσματα η έκθεση είχε βασιστεί σε μια έκθεση του ΚΟΠΑΘΕ του 2007. Δεν υπήρχε χρόνος να ε, ληφθούν ε, πιο πρόσφατα στοιχεία και η έκθεση αυτή του 2007 βαζόταν σε στοιχεία του 2005. Ήταν λοιπόν κάπως παροχημένα όλα αυτά η ανάλυση για τους σπόρους λοιπόν, για τους αλευτικούς σπόρους. Και δεν είχε ληφθεί υπόψη και η τελευταία ανάλυση που είχε κάνει η μεικτή επιστημονική επιτροπή που είχε δημιουργηθεί στα πλαίσια της συμφωνίας. Δεν είχαν λοιπόν εκτιμηθεί σωστά τα δεδομένα. Τώρα λοιπόν που έχουμε ε, όλα αυτά τα στοιχεία μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα. Και ε, η πολιτική για τον αλληλευτικό κλάδο. Το παλιό πρωτόκολλο ήταν πολύ αναλυτικό για το πώς έπρεπε να εφαρμοστεί η πολιτική και οι χρηματοδοτήσει στον τομέα αυτό και χρειάστηκε πολύς χρόνος για να ξεκινήσει η χορήγηση αυτών των πιστώσεων προς τον κλάδο. Μέχρι να μπορέσουν να συνεδριάσουν κάποιες μικρές επιτροπές για να ε, συμπεριληφθούν όλα αυτά στην συνολική στρατηγική και τώρα έχουν αρχίσει να λειτουργούν καλύτερα όλα αυτά. Με βάση αυτές τις επικρίσεις και έχοντας ακούσει τι είπε και ο κύριος Διευθυντής, πώς αυτά τα τρία θέματα, οικονομικό, κλαδικό, περιβαλλοντικό, πώς αντιμετωπίστηκαν, πώς κατά τη γνώμη μου αντιμετωπίστηκαν θετικά σε αυτό το νέο πρωτόκολλο, πώς επιλύθηκαν. Το οικονομικό. Δεν θα επαναλάβω τώρα όλα τα στοιχεία, αλλά ορισμένα στοιχεία πρέπει να τα πω. Ότι παρά το ότι ο αριθμός σκαφών μειώθηκε από 137 σε 126, οι δυνατότητες αλίευσης, όπως είπε ο κύριος Ντεπίπερ, αυξήθηκαν κατά 33%. Κυρίως λόγω της κατηγορίας 6 που είναι τα πελαγικά παραγαδιάρικα. Εάν δούμε συνολικά όχι μόνο το κόστος για τον κοινωτικό προϋπολογισμό, και αλλά, και το τμήμα των εφοπλιστών. Το σύνολο του κόστους έχει αυξηθεί μόνο κατά 1% λαμβάνοντας τι πληρώνουν, υπόψη τι, λαμβάν, τι πληρώνουν και οι εφοπλιστές. Αυτό λοιπόν που πρέπει να τονίσουμε και που είναι σημαντικό είναι, είναι ότι το βάρος για τον ενωσιακό προϋπολογισμό μειούται κατά 17% από 36,1 εκατομμύρια περνάει στα 30 εκατομμύρια. Επαναλαμβάνω λοιπόν, για τον προπολογισμό της Ένωσης ε, έχουμε μείωση 17% του κόστους. Και καλύπτεται από την αύξηση της ε, συνεισφοράς των εφοπλιστών. Στο προηγούμενο πρωτόκολλο πλήρωναν 3,4 εκατομμύρια, τώρα οι εφοπλιστές θα πληρώσουν 10 εκατομμύρια. Όπως θα θυμάστε, σε σχέση με την έκθεση ex post, όπου ελέγεται ότι η σχέση κόστους ε, ένωσης, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης εφοπλιστών ήταν 9% για την Ένωση και 9% για τους εφοπλιστές, τώρα είναι 75% για την Ένωση και 25% για τους εφοπλιστές και αν λάβουμε υπόψη το σύνολο της συμφωνίας και αν λάβουμε υπόψη μόνο την εμπορική συμφωνία, αυτό που πληρώνει δηλαδή για το δικαίωμα αλληλείας, εδώ υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση. Η σχέση γίνεται 62 ένωση 38 εφοπλιστές. Οπότε, πάνω κάτω, το ποσό είναι το ίδιο, αλλά η σύστασή του ε, είναι διαφορετική, συμμετέχουν πολύ περισσότερο εφοπλιστές, ε, όπως ε, είπαν πολλοί, έχει να κάνει με την μεταρρύθμιση, έχει να κάνει με τις νέες συμφωνίες αλίας, όπου γενικά έχει ζητηθεί να ε, συμβάλλουν περισσότερο και καλύτερα εφοπλιστές. Επίσης, όπως είπε ο κύριος Ντεπίπερ, επειδή επιλύθηκε ένα από τα σοβαρά προβλήματα που είχαμε επισημάνει ότι τα, μετρικά, τεχνικά μέτρα για ορισμένες κατηγορίες αλίες δεν τα κατάλληλα. Δηλαδή υπήρχαν οι δυνατότητες αλλά τα τεχνικά ε, μέτρα δεν ήταν τα κατάλληλα και γι' αυτό ορισμένες κατηγορίες όπως οι 4 δεν είχαν μπορέσει πλήρως να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Και είχε υπάρξει λοιπόν υποχρησιμοποίηση. Κυρίως για την κατηγορία 4 που είχε χρησιμοποιηθεί πολύ λίγο γιατί τα τεχνικά μέτρα για τα σκάφη και τα λοιπά δεν ήταν τα κατάλληλα, σε αυτό το νέο πρωτόκολλο όλα αυτά έχουν ξεπεραστεί. Αυτή η υποχρησιμοποίηση για ορισμένες κατηγορίες δεν θα πρέπει λοιπόν τώρα να σημειωθεί. Περιβάλλον. Ειλικρινά σας λέω, και εδώ ακόμη περιμένω κάποια στοιχεία που ζητήσαμε από το Μαρόκο. Ακόμη τα περιμένω συγκεκριμένα στοιχεία για να έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Αλλά γενικά πιστεύω ότι οι συμβαλόμενοι και το Μαρόκο δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι επιστήμονες που συμμετείχαν στις συνεδριάσεις για τον υπολογισμό των πλεονασμάτων και οι εθνικές διοικήσεις όλοι λοιπόν συμφωνούν ότι οι μελέτες που μας υπέβαλαν οι μαροκινοί επιστήμονες ήταν σοβαρές και πλήρεις σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων εξηγώντας, αποτιμώντας με βάση τις δυνατότητες αλίας που ε, υπήρχαν. Θα σας πω λοιπόν στη συνέχεια πιο συγκεκριμένα πράγματα αλλά ε, πρέπει να σας πω ότι το Μαρόκο ε, είχε, ε, το Μαρόκο απέρριψε τις 100.000 τόνους που είχαμε ζητήσει για τα ε, βενθοπελαγικά είδη. Δέχθηκαν μόνο 80.000. Και για το Μαρόκο επίσης απορρίφθηκε μια νέα αίτηση. Είπε το Μαρόκο ότι δεν μπορεί να εγκρίνουν νέες κατηγορίες αλίας. Τις απέρριψαν. Επίσης απέρριψε το Μαρόκο την δυνατότητα παράπλευρων αλλιευμάτων σε κεφαλόποδα, σε ε, καρχαρίες και σε οστρακοειδή. Και σε, όχι σε, κεφαλ, ε, σε μαλάκια, όχι οστρακοειδή. Έχουμε σοβαρά λοιπόν επιστημονικά στοιχεία που μας υποβλήθηκαν στους τους Μαροκινούς για να απορριφθούν ορισμένα από τα αιτήματά μας. Επιπλέον, Υπάρχει ένα στοιχείο ελέγχου που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Έχω συμμετάσχει σε διάφορες μικτές επιτροπές και είδα επανειλημμένα τις διαμαρτυρίες των Μαροκινών για το ότι τα στοιχεία που ελάμβανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν ακριβή. Τώρα έχουμε το παράρτημα 11 που θέλει να δημιουργήσει ένα σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής όλων των αναγκαίων πληροφοριών. Δηλαδή έχει ξεκινήσει η διαδικασία η ανταλλαγή να γίνεται με ηλεκτρονικό, σοβαρό και τελειωτικό τρόπο για να μην υπάρχουν πλέον στο μέλλον καθόλου διαμαρτυρίες. Έχουμε λοιπόν τις αναγκαίες μεθόδους που νομίζουμε ότι είναι ιδιαίτερα σκόπιμες. Όλα αυτά αναφέρονται στο παράρτημα 11 και στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αναφέρεται ότι θα υπάρχει πολύ σοβαρή επιστημονική προσπάθεια συντονισμού. Έχουν δεσμευτεί δηλαδή οι πλευρές να έχουν τακτικά, όχι όπως το παρελθόν που καμιά φορά όταν μας ζητούσαν ότι θα υπάρχει τακτική, τακτική επαφή, τακτικές επιστημονικές συνεδριάσεις για να επιλύονται τα επιστημονικά θέματα που μπορεί να θέσει οποιαδήποτε μεικτή επιτροπή. Αυτό ο μόνιμος λοιπόν χαρακτήρα είναι αυτός που καθιστά πολύ σοβαρότερη την επιστημονική συνεργασία, τον επιστημονικό συντονισμό. Είπε ο κύριος Δεπίπερ ότι το Εθνικό Ινστιτούτο ε, ε, ε, Αλλιευτικών Μελετών του Μαρόκου είναι πολύ σοβαρό και εγώ το επισκέφτηκα. Ασχολούνται 300 επιστήμονες εκεί. Είναι σημαντικό λοιπόν ίδρυμα, ε, έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα οι δραστηριότητες έρευνας που κάνει. Συνολικά λοιπόν έχουμε εγγυήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, για τους ελέγχους, για την μόνιμη επιστημονική παρακολούθηση καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του πρωτοκόλου. Και για τον κλάδο τώρα γενικά, για τον τομέα της αλίας. όπου είχε ζητηθεί περισσότερη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο. Γιατί κάποιες νομικές εκθέσεις είχαν διαμαρτυρηθεί γι' αυτό. Και εδώ έχουμε τώρα πρόσφατα στοιχεία, ή μάλλον μας λείπουν κάποια πρόσφατα στοιχεία, αλλά στο νέο άρθρο 6 συμμορφούνται πλήρως με αυτό που είχε απαιτήσει το Κοινοβούλιο και η ε, εντολή του Συμβουλίου που περιέχει πολύ σαφείς κατευθυντήριες γραμμές προς την Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις. Και συγκεκριμένα εκεί αναφέρεται και η διεθνής νομιμότητα. Στο νέο άρθρο 6, που είναι απόλυτα καινοτόμο, συμμορφούνται το πρωτόκολλο, σε αυτά που είπα προηγουμένως, για τη χρήση από το Μαρόκο της οικονομικής αντιστάθμισης για τη στήριξη του τομέα. Ούτως ώστε να ωφεληθεί ο τοπικός πληθυσμός. Το Μαρόκο θα ενημερώνει τακτικά για τα οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη για τον πληθυσμό από πλευράς απασχόλησης, επενδύσεων και άλλων μετρησίμων επιπτώσεων και για την γεωγραφική κατανομή όλων αυτών των ωφελημάτων. Από εδώ και εφ' εξής, όπως αποδέχθηκε το Μαρόκο, θα πρέπει να μας δίνουν και κατά περιφέρειες πόσες επενδύσεις έχουν γίνει, πόσες θέσεις εργασίας έχουν ε, διαπιστωθεί κτλ. Αυτό είναι καινούργιο στοιχείο, καινούργιο στοιχείο, πρώτη φορά το βλέπω σε ένα τέτοιο πρωτόκολλο. Αυτό ανταποκρίνεται στα αιτήματα που έχουμε υποβάλει και ως Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οπότε θεωρώ ότι αυτά ήταν τα τρία στοιχεία κλειδί για την απόρριψη του προηγούμενου πρωτοκόλου, οπότε τα θέματα αυτά έχουν επιληθεί στο νέο πρωτόκολλο. Λοιπόν, τώρα για τη διαδικασία, για το πώς τα πληρώματα για πρώτη φορά θα ε, νιολογούνται, θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο κατάλογος, ένα, νιολο, ένα δηλαδή ε, ένας κατάλογος, ένα μητρό με τις ιδιότητές τους γιατί ξέραμε ότι ε, στο παρελθόν ε, τα πληρώματα άρχισαν, μπάρκαραν χωρίς να έχουν καμία προηγούμενη εκπαίδευση. Θα υπάρχει ένα μητρό λοιπόν που θα αναφέρεται ποιοι μπαρκάρουν, τι προσόντα έχουν. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και αυτό καινούριο στοιχείο. Κάτι άλλο σημαντικό που είχε στήσει στο Μαρόκο ήταν το θέμα των εκφορτώσεων λήφθηκε υπόψη και από τις δύο πλευρές. Γιατί και το Μαρόκο έκανε μια προσπάθεια για να επεκταθούν οι δυνατότητες εκφόρτωσης για να συμπεριληφθούν και ορισμένα ε, λιμάνια που έχουν την αναγκαία υποδομή. Όπως για παράδειγμα το λιμάνι στο Μοχαμεντία που είναι πολύ καλύτερο από ορισμένα που προβλέπονταν προηγουμένως. Όπου τα σκάφη είχαν πρόβλημα για να κάνουν την εκφόρτωση. Όπως διαπιστώνεται λοιπόν λήφθηκαν υπόψη πολλά θέματα. Νομίζω ότι το πιο θετικό στοιχείο από την απόρριψη της προηγούμενης ε, συμφωνίας του 2011, του προηγούμενου πρωτοκόλλου, της παράτασης του προηγούμενου πρωτοκόλλου, βεβαίως έκανε μεγάλη ζημιά σε πολλά σκάφη, δημιούργησε πολλά οικονομικά πρόβληματα για πολλούς, αλλά είχε το θετικό στοιχείο ότι οι επικρίσεις που είχαμε τότε διατυπώσει λήφθηκαν υπόψη και από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή κατά τις διαπραγματεύσεις και βεβαίως και από πλευράς του Μαρόκου. Και συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Ντεπίπερ, αυτό το νέο πρωτόκολλο έλαβε υπόψη όλα μας τα αιτήματα Γενικά βέβαια υπάρχουν λεπτομέρειες που θα μπορούσαν ακόμη να βελτιωθούν και θα βελτιωθούν ε, μέσω των συνεδριάσεων των μεικτών επιτροπών στη συνέχεια, αλλά συνολικά νομίζω ότι η αποτίμηση που θα πρέπει να κάνουμε είναι θετική. Ε, με συγχωρείτε που μίλησα και διαδικασία, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να τα αναφέρω αυτά. Ε, με συγχωρείτε που μακρηγόρησα. Ευχαριστούμε κύριε κυρία Φράγκα επειδή είστε εισηγήτρια, ήταν πολύ σημαντική αυτή η παρουσίαση. Έχω 10 αγορητέ και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μα. Θα παρακαλούσα να, γίνει, να είστε όσο πιο σύντομοι γίνεται. Κύριε Ρομέδα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω μόνο ορισμένε παρατηρήσει αλλά και κάποιε ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά κύριο λόγο. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη μου παρατήρηση έχει να κάνει με ένα από τα βασικά ζητήματα που ήδη υπήρχε και στο παρόν πρωτόκολλο. Πρώτα απ' όλα ε, πρόκειται για την ασάφεια δηλαδή του γεωγραφικού πεδίου, της γεωγραφικής κάλυψης. Θα έπρεπε να μας καθησυχάζετε και εδώ στο Κοινοβούλιο. Τέσσερις από έξι περιοχές στην, στα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας ε, δεν έχουν απαγόρευση για αλία. Εδώ όμω υπάρχει ένα θέμα ορισμών πρέπει να υπάρξει καλύτερος ορισμός. Επίσης, μιλάμε για τα ύδατα που εμπίπτουν εντό της κυριαρχίας του βασιλείου του Μαρόκου. Από νομικής πλευράς, εάν το ερμηνεύσουμε, αυτό σημαίνει ότι αποκλείονται τα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας. Αν όμως βασιστούμε σε προηγούμενες εμπειρίες μας και στο ότι έχουμε μάθει από το παρελθόν, συνειδητοποιούμε ότι ο αποκλεισμό αυτός δεν είναι πραγματικός μάλιστα ε, ό,τι δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Βασιλείου του Μαρόκου ε, μπορεί να χρησιμοποιείται σαν να ήταν στη δικαιοδοσία τους, αντίθετα με το διεθνές δίκαιο. Κάτι άλλο που είναι επίσης ενδιαφέρον είναι η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει ένα νέο τμήμα κειμένου για τις ευθύνες εκπλήρωσης αρχών και υποχρεώσεων σε σχέση με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί δεν υπάρχει κάτι τελείως καινούριο. Η μνή αυτή υπήρχε και στο προηγούμενο πρωτόκολλο. Αλλά αυτό δεν άλλαξε και πολλά ως προς την ε, εκτέλεση του πρωτοκόλλου. Οπότε ούτω ή άλλω δεν μου φαίνεται ακριβή η διατύπωση. Για το οικονομικό τώρα σκέλο, ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκε, ώστε να μην προχωρήσει. Να μην παραταθεί το ισχυρό πρωτόκολλο. Και αυτό χρήζει συζήτηση. Ακούσαμε μεγάλη προσοχή όσα είπε η συνάδελφος Κάρμεν Φράγκα για την εκπόνηση της μελέτης που έγινε για να υπολογιστεί η αναλογία κόστους ωφελία. αλλά η κατάσταση αυτή έχει μειώσει τα κονδύλια θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια έξοδα θα τα καλύψει ο ίδιο ο τομέα. Το ερώτημα όμω είναι πώ αυτέ οι επενδύσει θα αξιοποιηθούν. Ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω γενικά την Επιτροπή να μα πει εάν υπάρχει νέα μελέτη, εξάντε μελέτη για το κόστο και την ωφέλεια. Έχετε κάνει κάτι εκ των προτέρων για να δούμε από οικονομικής πλευρά ποιε είναι οι προβλέψεις. Διότι ακόμη και με τα σημερινά νούμερα είναι ασαφές για τη γεωγραφική κατανομή τώρα. Και πάλι, λυπάμαι που το λέω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει σε μία και μόνο πτυχή. Ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο καλύπτονται τα ωφέλη του τοπικού, ε, τα, τα συμφέροντα του τοπικού πληθυσμού. Να θυμίσω τα εξή δύο στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, το νομικό πλαίσιο μιλά και για τις επιθυμίες όχι μόνο του τοπικού πληθυσμού, αλλά των ανθρώπων της χώρας. Αυτό είναι ελαφρώς διαφορετικό. Και δεν καλύπτεται αυτό από την έκθεσή σας. Και επί τη ουσία αυτό που δεν περιλαμβάνει αυτή η έκθεση είναι κάτι ζωτική σημασία κατά την άποψή μου. Διαβουλεύσει με του ανθρώπου τη χώρα. Κανεί δεν του ρώτησε τη γνώμη του. Κανεί δεν ρώτησε του ανθρώπου τη Δυτική Σαχάρα τι θέλουν. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία εγγύηση ότι θα συμμετάσχουν όντω στην όλη διαδικασία. Και για να ολοκληρώσω τις την παρέμβασή μου, για τους ε, ψαράδες από το Μαρόκο και τη συμμετοχή τους. Πώς ξέρουμε ότι οι... τους ναυτιλωμένους δεν θα συμπεριλαμβάνονται και αλείς από τη Σαχάρα. Πώς ξέρουμε ότι θα γίνει αυτό και ότι θα μπορέσουν να αποφεληθούν από τη συμφωνία. Για το μηχανισμό παρακολούθησης και ελέγχου επίση έχω κάποιες παρατηρήσεις, αλλά είναι πιο τεχνικές. Να ολοκληρώσω με δύο παρατηρήσεις. Για, την, ε, για τις απορρίψεις των αλλιευμάτων, μάλλον για τι εκφορτώσεις των αλλιευμάτων. Η υποχρέωση αλλίευση γάδου σε ελεύθερα ύδατα μπορεί να θεωρηθεί ως μια συνεισφορά στην νόμιμη μηχανία ελίας. Σε αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφεί. Πρέπει να έχουμε πλήρη συνέστηση για να μην αντιμετωπίσουμε κάτι που μπορεί να δημιουργήσει άλλε ανησυχίε. Και τέλο, αυτή είναι η ακροτελεύτια παρατήρησή μου. Ω προ την περιβαλλοντική κατάσταση, το, πώς, ε, το τι συμβαίνει εκεί με του πόρου, του ελευτικού πόρου. Θα ήθελα να γνωρίζουμε πώ κάνατε του υπολογισμού σα. Πώς, πώς μετρήσατε την κατάσταση των αλλιευμάτων εκεί. Θέλουμε μια ε, αυστηρή, ακριβή ε, αποτίμηση για να μπορέσουμε να πάρουμε την απόφασή μας. Αλλά με τη σημερινή κατάσταση, αν αυτό δεν το δούμε μπροστά μας, θα είναι πολύ πρόημο να εγκρίνουμε την έκθεση αυτή. Ευχαριστούμε κυρία Πατράου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι πραγματικά συνοπτική διότι μετά την εισηγήτρια Κάρμεν Φράγκα και την παρουσίασή της, ε, πραγματικά καλύφθηκα. Δεν θα επαναλάβω όσα είπε. Θα ήθελα σε μια πρώτη φάση να επιστήσω την προσοχή σας και νομίζω ότι αυτό είναι το πλέον σημαντικό ότι χάθηκαν πολλά από αυτά που είχε καταψηφίσει το Κοινοβούλιο προς αυτή τη συμφωνία. Όχι απλώς χάθηκε ό,τι είχε να κάνει με τις αλληλευτικές δυνατότητες, αλλά και ό,τι είχε να κάνει με τις ευρύτερες πολιτικές ισορροπίας και τις ε, πολιτικές σχέσεις με τις ε, όμορες χώρες. Ξέρουμε ότι η γεωγραφική θέση του Μαρόκου είναι εξαιρετικά σημαντική, ιδίως για τις χώρες του Νότου. Αυτό λοιπόν που στο παρελθόν είχε να κάνει με την έγκριση της συμφωνίας και την καθόρισε δεν ήταν μόνο ο τομέας της αλίας αλλά οι σχέσεις μας με μια χώρα που είναι και γειτονική. Πέραν του γεγονότος ότι χάσαμε πολλά από τον τομέα της αλίας ούτως ή άλλως αλλά τώρα αν έχουμε 727 σκάφη, αν οι ελληνικές προσπάθειες είναι μεγαλύτερες παρά την αντίθετη διάθεσή μας, να θυμίσω ότι ούτως έλος και πριν είχαμε 800 σκάφη στα νερά του Μαρόκου. Δεν είναι ότι χάσαμε ε, τη γη κατά τα πόδια μας ή το νερό τέλο πάντων για να είμαστε και στο ανάλογο πλαίσιο. Όμως τα επικριτικά σχόλια που διατυπώθηκαν στο παρελθόν σε σχέση με το πρωτόκολλο που καταψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο Αυτά τα επικριτικά σχόλια θα ήθελα να είχαν ε, ληφθεί υπόψη σοβαρά και να υπήρχαν και αποκρίσεις αυτές τις επικρίσεις. Όπως είπε και η Κάρμεν, βεβαίως περιθώριο για βελτιώσεις υπήρχε. Αλλά ότι στις επικρίσεις του Κοινοβουλίου ε, υπήρξε ήδη κάποια ανταπόκριση. Αυτό έγινε. Και ότι η έκθεση αντικατοπτρίζει κάποιες από τις θέσεις μας και αυτό ισχύει. Και να θυμίσω και κάτι άλλο, κάποιες προοπτικές που πάντοτε πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν μιλάμε για πρωτόκολλα και αλλιευτικές συμφωνίες. Πρώτα απ' όλα η πολιτική διάσταση που έχει να κάνει με την παρουσία μας στα τα τρίτων χωρών. Γνωρίζουμε άψογα ότι όπου δεν πάμε εμείς ε, θα καλύψουν τη θέση μας άλλοι, με ανάλογες διαθέσεις όπως εμείς. Στο Μαρόκο είναι σημαντικό να έχουμε μια παρουσία. 1% βέβαια είναι η παρουσία μας, δεν είναι και τίποτα φοβερό, αλλά είναι σημαντική για μα. Η πολιτική διάσταση πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη. Είναι η παρουσία μα στα διεθνή ύδατα, στον κόσμο. Μία ε, παρουσία η οποία πρέπει να συνδυάζεται με πολλά κριτήρια ευθύνη και σε περιβαλλοντικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Και το οικονομικό σκέλο. Η συμφωνία αυτή είναι ουσιαστική σημασία για το στόλο μα. Είναι από τι πλέον σημαντικέ συμφωνίε για του στόλου τη Ευρώπη από την οικονομική οπτική γωνία. Εδώ λοιπόν έχουμε μία νέα συμφωνία με αύξηση 25% του κόστους για τους ίδιους τους πλειοκτήτες. Η πρόταση λοιπόν αυτής συμφωνίας δείχνει ότι αυτή η αύξηση του κόστους δεν τους εμποδίζει να θέλουν να τονίσουν την παρουσία τους σε αυτή την περιοχή. Για πολιτική διάσταση και την οικονομική μίλησα, ας σταθώ τώρα και στα κοινωνικά. Ως προς το κοινωνικό σκέλος υπάρχει σαφής βελτίωση, να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή δηλαδή στα κοινωνικά δικαιώματα, προκειμένου να εφοληθούν και οι Μαροκινοί από την παρουσία μα στα υδατά του. Και τελευταίο σημείο, γιατί υποσχέθηκα να είμαι σύντομη, ε, το είχα υποσχεθεί μόλις ξεκίνησα, ε, περιβαλλοντικό ε, σκέλος. Και εδώ υπάρχει ενδυνάμωση σε αυτό το σχέδιο πρωτοκόλλου. Να ολοκληρώσω λέγοντα ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρωτόκολλο που κατά πάσα πιθανότητα είναι το πλέον ακριβέ ε, και ε, αυστηρό και συγκεκριμένο αλλά και φιλόδοξο που ω τώρα έχουμε δει στην Επιτροπή Αλίας. Εύχομαι να ακολουθήσουν και άλλα. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλα. Όμως έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια, υπήρξαν ε, ικανοποιητικές απαντήσεις και γενικώ μεγάλες προσδοκίες και απαιτήσει. Αυτή είναι η πλέον λοιπόν ικανοποιητική πρόταση με πολύ μεγάλες απαιτήσει που πέρασε από τα χέρια μας. Σήμερα οι άλλες τρεις συμφωνίες που εξετάζουμε δεν είναι αυτού του επίπεδου. Θέλω λοιπόν να επαναλάβω με μεγάλη σαφήνεια την απόλυτη στήριξή μου στη συμφωνία αυτή όπως μας έχει υποβληθεί και να ευχαριστήσω θερμά την Κάρμεν Φράγκα για την τόσο διεξοδική ανάλυση των διαφόρων σημείων αυτής της συμφωνίας που ακριβώς αιτιολογούν και τη στήριξη μου. Ευχαριστώ. Thanks Ευχαριστώ πολύ, ε, Ευχαριστώ. Για να είμαι σύντομο, θα σταθώ σε ένα και μόνο από τα σημεία που μας δυσκόλεψαν και είχαν ε, σταθεί αιτία για την προηγούμενη καταψήφιση του πρωτοκόλλου από το Κοινοβούλιο. Κάτι που έχει απασχολήσει την Επιτροπή μα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οικονομική λόγοι, περιβαλλοντική, κοινωνική. κάτι ακόμη που είχε θερε... και ένα ακόμη σημείο που είχε θεωρηθεί παραβίαση του διεθνού δικαίου. Και εγώ σε αυτό το τελευταίο θα σταθώ. Ε, δεν συμφωνώ απολύτω με το ΣΕΠΕ συνάδελφο Παντραού ότι η μη έγκριση του πρωτοκόλλου στο παρελθόν ε, ζημίωσε τον Ευρωπαϊκό Στόλο και το Μαρόκο. Τι μπορούμε να κάνουμε ε, για τις ζημιές αυτές δεν μπορούμε να εγκρίνουμε μια παράνομη συμφωνία που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πολλές ευκαιρίες ε, ανά τα χρόνια για να διορθώσει, να βελτιώσει τη συμφωνία και να την ευθυγραμμίσει με το διεθνέ δίκαιο. Δεν το έκανε. Εμεί επιστήσαμε την προσοχή σα επανειλημμένω για αυτή την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν άλλαξε στάση. Αυτό είναι κάτι που μπορούσε να συμβεί και προφανώ συνέβη. Είχαμε και την καταψήφιση και υπήρχαν ζημιέ για του τόλου πολλών χωρών. Γι' αυτό θα έπρεπε να αναλάβει ευθύνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι προτάσει έχουμε τώρα μπροστά μα. Μια πρόταση που υπό την άποψη αυτή και σε σχέση με τις ανησυχίες μας για το διεθνές δίκαιο σε τίποτε δεν διαφέρει από την προηγούμενη. Δηλαδή, εάν η προηγούμενη συμφωνία επέτρεπε την αλία σε είδατα που βάσει του διεθνούς δικαίου δεν ανήκουν στην, κυριαρχία, στην δικαιοδοσία του Μαρόκου, η νέα πρόταση τι προτείνει ακριβώς τη συνέχιση της προηγούμενης κατάστασης. Θα έπρεπε να οριστεί με σαφήνεια, η συμφωνία θα έπρεπε να ορίζει με σαφήνεια ποια είναι τα εθνικά ύδατα του Μαρόκου, αποκλείοντας τα ύδατα του, ε, της Σαχάρας ε, και της Μεσογείου, αλλά και του Μεσημβρινού 2740. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η αυλεψία να μην αγνοηθεί από πλευρά μα. Είναι παραβίαση του διεθνού δικαίου. Και το είπε και το ποινικό δικαστήριο τη Χάγη. Δεν αναγνωρίζει την εθνική κυριαρχία του Μαρόκου στα είδατα αυτά. Έχουμε λοιπόν μπροστά μα μια συμφωνία που επιτρέπει την αλεία. Μια συμφωνία με ένα κράτο όπω το Μαρόκο. Λοιπόν, επιτρέπεται συμφωνία σε ύδατα που το διεθνέ δίκαιο έχει καθορίσει ότι δεν είναι στην ε, δικαιοδοσία του Βασιλείου του Μαρόκου. Ε, δεν είναι αυτό παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αυτό πρέπει να διορθωθεί και ελπίζω να διορθωθεί. Να αποκλειστούν τα ύδατα που βρίσκονται νοτίως του Μεσοβρινού 2740. Μιλάμε για εθνικά ύδατα της Δυτικής Σαχάρας που υπό την έννοια του διεθνούς δικαίου δεν ανήκουν στο Μαρόκο. Δεν μπορούμε λοιπόν να θεωρούμε ηθική μια τέτοια συμφωνία. Να θυμίσω επίση ότι οι αντιρρήσει μα ε, ω προ αυτό το θέμα ε, είχαν να κάνουν ε, και με την άρνηση του Κοινοβουλίου με νομικά έτη, νομική βάση. Δηλαδή, θυμήσαμε τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για τα εθνικά είδατα του Μαρόκου. Το δικαίωμα των κατεχόμενων επίσης ε, λαών, ε, να, εδαφών, των ανθρώπων των κατεχόμενων εδαφών, να εκμεταλλεύονται τους φυσικούς πόρους των περιοχών τους. Αυτό αφορούσαν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε για μια διάταξη ανάλογη με αυτή που ε, ανέφερε η εισηγήτρια και συμπεριλαμβάνεται στο τωρινό πρωτόκολλο. Οι μαροκινές αρχές Εφ' εξής, θα πρέπει να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατανομή των ωφελών σε ε, δαφικό επίπεδο και τη γεωγραφική κατανομή θα πρέπει να την εξηγούν λεπτομερώς και αν αυτό δεν επιληθεί ως πρόβλημα έχει να κάνει η όλη κατάσταση με τα δικαιώματα του λαού της Σαχάρας και με το πώς εκμεταλλεύονται τους φυσικούς τους πόρους και τα ψηφίσματα του ΙΕΠ προανέφερα. Το ευρωπαϊκό δίκαιο και το διεθνώς, διεθνές δίκαιο ε, ε, επιβάλλει, αυτά να, να ληφθούν υπόψη. Είναι βασικότατο αυτό. Δεν ε, άκουσα τι έκανε εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχε δύο επιλογές. Η καλύτερη ήταν απλά και εξάστερα να αποκλείσει τα ύδατα αυτά από το πεδίο της συμφωνίας ή έστω να ακούσει τους εκπροσώπους της Δυτικής Σαχάρας, των ανθρώπων της Δυτικής Σαχάρας. Είναι γνωστοί, υπάρχουν διαπραγματεύσεις εδώ και χρόνια στο επίπεδο του ΑΕΜ με αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν ήρθαν οι νόμιμοι αυτοί οι εκπρόσωποι των ε, Σαχαριανών να μιλήσουν και να εκφραστούν για αυτή τη συμφωνία. Αυτό διακυβεύει την βασική αρχή που ήδη είχαμε επικαλεστεί ε, στη νομική μας νομοδότηση ως Κοινοβούλιο. Την είχαν ετοιμάσει οι νομικές μας υπηρεσίες για την προηγούμενη μορφή της συμφωνίας. Και ακριβώ με τον ίδιο τρόπο ε, η γνωμοδότηση αυτή θεωρούσε ότι δεν καλύπτονταν οι προποθέσει για να θεωρηθεί η συμφωνία νόμιμη. Θα καλύπτονταν ε, οι περιπτώσεις αλίευσης από κάποια σκάφη στα έδατα της Δυτικής Σαχάρας με τη συμφωνία όπως είχε διατυπωθεί στο παρελθόν. Άρα αυτό το πρόβλημα από νομική πλευράς για μας παραμένει. Δεν έκανε τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το λύσει. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι όλοι, όλοι οι συνάδελφοι εδώ προφανώς θέλουν η συμφωνία να ε, προχωρήσει και να ε, κυρωθεί. Όμως, εάν μια από τις χώρες σας κατεχόταν από ξένη δύναμη, με το ίδιο βλέμμα θα αντιμετωπίζετε αυτή τη, θα βλέπατε αυτή τη συμφωνία, θα αφήνατε στους, ε, στις δυνάμεις κατοχής να εκμεταλλεύονταν ενόχλητοι τους φυσικούς σας πόρους. Μιλάμε για πόρους, των οποίων την, ε, τους οποίους θα έπρεπε να ε, καρπώνονται οι άνθρωποι της χώρας, του, της περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι έλυσε το πρόβλημα. Όχι, θα μπορούσε να το λύσει πολύ, με πολύ απλό τρόπο, εάν απέκλειε τα τα νοτίως του Μεσημπρινού 2740. Ή έστω ακούγοντα του εκπροσώπου του λαού τη Δυτική Σαχάρα, για να πούν και αυτή την άποψή του για αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Συγνιού. Ε, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα ανοιχτό μικρόφωνο από έναν συνάδελφο. Ευχαριστώ που το κλείσατε. Λοιπόν, δεν θα πω ότι θα είμαι σύντομο, γιατί κάθε φορά που το λέμε αυτό είναι ένα κωδική ονομασία του θα μιλήσω 10 λεπτά. Λοιπόν, αναφερόμαστε στο δικαίωμά μα να συνεχίσουμε την αλληλεία στα ύδατα του Μαρόκου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη ανέφερε ότι η αύξηση θα είναι τη του 33% και αυτό αφορά κυρίως τους βιομηχανικούς ε, στόλους. Ποιο θα είναι ο κόστος για τους ε, φορολογούμενους, ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ και αυτό δυσανάλογα θα το επιμιστούν οι Βρετανοί φορολογούμενοι. Γιατί φυσικά τα περισσότερα από αυτά τα αλλιευτικά για τα οποία μιλάμε προέρχονται από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι αυτή είναι μια μορφή βοήθειας ε, προς τρίτη χώρα. Ε, αναρωτιέμαι όμως, εάν θα είχα τη δυνατότητα να αξιολογήσω εάν τα χρήματα του Βρετανού φορολογούμενου χρησιμοποιούνται προς σωστούς σκοπούς και αν θα έχω τη δυνατότητα να πάω στο Μαρόκο και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το αξιολογήσω αυτό. Για φανταστείτε λοιπόν ότι αυτά τα λευτικά από την Ισπανία και την Πορτογαλία μπορούν να πάνε στην ανοιχτή θάλασσα, να αλλιεύσουν, μετά να τα μεταφορτώσουν σε μια μικρότερη, στο μικρότερο στόλο των Μαροκινών και αυτά να ε, εξαχθούν στην ξηρά. Τελικά αυτό ποιον εξυπηρετεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να εστιάσω σε δύο στοιχεία. Πρώτον, το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ρήτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο συζητήτρια αρμόδια για την εξωτερική διάσταση της ε, πολιτικής αλίας. Προφανώς παρακολουθώ τη θέση του Κοινοβουλίου για αυτό το ζήτημα εδώ και καιρό. Πρώτη φορά που αποκτήσαμε μια ε, ουσιαστική θέση επ' αυτού του θέματος ήταν όταν ε, έγινε το κοινό ψήφισμα για την μελλοντική πρωτόκολλο με τη Μαυριτανία. Το 2011 ήδη είχαμε πει ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μια ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις συμφωνίες αλληλείας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών και οι οποίες θα πρέπει να ε, έχουν πριν από τις οποίες θα πρέπει να έχει προηγηθεί ένας ευρύς διάλογος με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών κοινοβουλίων. Αυτά το 2011. Μετά συμφωνήσαμε μια νέα κοινή πολιτική αλίας που συμπεριλαμβάνει ένα κεφάλαιο για την εξωτερική διάσταση, πολύ ξεκάθαρο. Αναφέρει ότι οποιαδήποτε συμφωνία βιώσιμη ε, για την αλλήλεια στο μέλλον θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μια ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ουσιαστικό στοιχείο της. Το Συμβούλιο συμφώνησε, επομένως υπάρχει η σύμφωνη γνώμη και των δύο συνομοθετών. Όταν λοιπόν το Συμβούλιο έδωσε την εντολή διαπραγμάτευσης για την Συμφωνία Λίας με το Μαρόκο, είπε το εξής και παραθέτω. Ακόμα και αν πρόκειται για εμπιστευτικέ πληροφορίε, όταν, όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινα δικαιώματα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είπε λοιπόν το Συμβούλιο ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ρήτρα που να προβλέπει τις συνέπειες σε περίπτωση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών αρχών. Αυτές ήταν οι εντολές του Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα και ήταν εξίσου σαφές ότι θα πρέπει να γίνεται σεβαστό το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι έχουμε λοιπόν εδώ στο νέο πρωτόκολλο. Μια εξαιρετικά ασαφή και νεφελώδη αναφορά που δεν είναι μια ρήτρα διακοπή τη εφαρμογή του πρωτοκόλλου σε περίπτωση παραβιάσεων των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Αυτό που λέει, αυτό που είναι στην πραγματικότητα είναι μια παραπομπή στην συμφωνία σύνδεσης που αναφέρεται στο διάλογο και στην ε, ενίσχυση της συνεργασίας. Αυτή λοιπόν η συμφωνία σύνδεσης λέει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών που καθιερώνει η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα πρέπει να εμπνέει τις ε, πολιτικές ε, και την ε, συνεργασία με το Μαρόκο. Επομένως κάνουμε μια παραπομπή σε μια άλλη συμφωνία η οποία με μεγάλη ασάφεια και πολύ γενικά λέει ότι απλώς θα πρέπει να εμπνεόμαστε από τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις αρχές και τις ρήτες ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουμε σε κάθε άλλη συμφωνία αλληλείας. Και για να πω και στην κυρία Πατράου Νίβας, εδώ πιστεύω ότι αυτό το πρωτόκολλο θα δημιουργήσει προηγούμενο. βρίσκεται στον αντίποδα οποιοδήποτε άλλου πρωτοκόλλου έχουμε συνάψει. Σε όλα τα άλλα πρωτόκολλα είναι μια, υπάρχει μια σαφής ρήτρα διακοπής ή αναστολής εφαρμογής του πρωτοκόλου. Αναφέρεται λοιπόν με σαφήνεια ότι ε, από τα, ε, σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα δύο μέρη παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχει δυνατότητα αναστολής του πρωτοκόλου ε, αλληλείας. Για παράδειγμα, συμφωνία με τη Γρυλανδία. Αναφέρεται σε αναστολή εάν υπάρχουν παραβιάσεις, και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως αυτές καταγράφονται όπως αυτά περιγράφονται μάλλον στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της Συμφωνίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, σε όλα τα άλλα πρωτόκολλα αναφερόμαστε σε αναστολή εφαρμογής του πρωτοκόλλου. Ειδικά για το Μορόκο, απλώς κάνουμε μια παραπομπή σε μια άλλη συμφωνία η οποία συμφωνία λέει ότι πρέπει να εμπνεόμαστε από τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το μόνο που λέει στην πραγματικότητα το πρωτόκολλο για το Μαρόκο είναι ότι σε περίπτωση σύγκρουσης διαφωνίας μπορεί να ανασταλεί η εφαρμογή του, χωρίς καμία αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και πιστεύω ότι εδώ έχει παραβιαστεί αυτό που συμφωνήσε το Συμβούλιο. Δεν έχει ακολουθηθεί η γνώμη του Κοινοβουλίου, ούτε η νέα κοινή πολιτική για την αλία. Ποια είναι λοιπόν τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορούν στο Μαρόκο, προφανώς το θέμα της Δυτικής Σαχάρας. Σας καλέσαν, να, κυρία συνάδελφε, να επισκεφτείτε το Μαρόκο. Εγώ προσπάθησα να επισκεφτώ τις κατεχόμενες περιοχές της Δυτικής Σαχάρας μαζί με τέσσερις συναδέλφους. Ε, τον προηγούμενο Υπουργό Εξωτερικών της Σλοβενίας, τον Όρμπετ Νόισερ, από τους σοσιαλιστές και, και άλλους. Ε, επίσης τον αναπληρωτή Γενικό ε, ε, Γραμματέα του ΟΗΕ πρώην. Ήταν ένας από τους συναδέλφους ο οποίος του σταμάτησαν στην Καζαμπλάνκα. Επιτροπή σας μιλάω. Η Επιτροπή με ακούει, αναρωτιέμαι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, αν ο κύριος Πίνο πρώην αναπληρωτής ε, γενικός γραμματέας του ΙΕ, τελευταία στιγμή αντιμετώπισε προβλήματα στην Καζαμπλάνκα, ήταν ένας από τους πέντε που προσπάθησε να επισκεφτεί τα κατεχόμενα εδάφη στην Δυτική Σαχάρα και τον σταμάτησαν και δεν είχε τη δυνατότητα να συναντήσει τους ανθρώπους εκεί. Αυτά συμβαίνουν και από την άλλη ε, ε, ε, εμείς είχαμε ενημερώσει τις αρχές του Μαρόκου, γνώριζαν ποιες είναι οι προθέσεις μας και προφανώς γι' αυτό μας σταμάτησαν. Εμείς θέλαμε να συζητήσουμε με τις αρχές του Μαρόκου, θέλαμε να συζητήσουμε με τις αρχές του Μαρόκου στην Δυτική Σαχάρα, αλλά δεν ήμασταν ευπρόσδεκτοι. Λάβαμε ένα, μια ε, ε, αγενέστατη επιστολή από τον ε, πρέσβη του Μαρόκο που μας ε, έλεγε ακτιβιστές. Μάλιστα. Απευθύνομαι λοιπόν στην Επιτροπή. Δεν μας επιτρέπουν να επισκεπτόμαστε την περιοχή εμάς γιατί είμαστε ακτιβιστές. Εσείς λοιπόν της Επιτροπής πώς καταφέρατε να επισκεφτείτε, να παρακολουθήσετε, να αξιολογήσετε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών στη Δυτική Σαχάρα. Πολύ θα ήθελα να μου απαντήσει η Επιτροπή. Πόσες φορές εκπρόσωποι της Επιτροπής μπόρεσαν να επισκεφτούν την περιοχή. Έχετε άραγε την πρόθεσμη, σι, να επισκεφτείτε την Δυτική Σαχάρα και να αξιολογήσετε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, η απάντηση την γνωρίζουμε. Καμία φορά εκπρόσωπος της Επιτροπής δεν επισκέφτηκε τη Δυτική Σαχάρα. Έχω φέρει εδώ ένα βιβλίο ε, από την Σουηδία, την ε, διοίκηση δύο Σουηδών δημοσιογράφων οι οποίοι προσπάθησαν να επισκεφτούν ε, και να καταγράψουν τι συμβαίνει εκεί και τους απέλασαν. Επομένω, τι συζητάμε για δημοκρατικές αρχές. Εσείς μας μιλάτε για την γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων και ούτε καν μια αναφορά στη Δυτική Σαχάρα δεν υπάρχει στο κείμενο της ε, Επιτροπής ε, Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και τη διεθνή κοινότητα πρόκειται για ένα, μια, μια περιοχή, μια εδαφική περιοχή η οποία δεν ασκεί ε, κυριαρχία. Πώς λοιπόν μπορούμε να επιτρέψουμε στα αλλιευτικά, τα ευρωπαϊκά, να αλλιεύουν σε μια περιοχή που δεν, ε, που δεν ανήκει σε κάποιο κράτος. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα νομιμότητας. Ρωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς προτίθεστε να παρακολουθείτε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα δάφη της Δυτικής Σαχάρας. Πρόκειται να, για παράδειγμα, στείλετε μια επίσημη αποστολή η οποία θα συναντηθεί με το Πολυσάριο που θα, θα επισκεφτεί τις φυλακές. Θα το τολμήσετε αυτό? Και αν όχι, αυτό δεν αποδεικνύει ότι αυτή η συμφωνία δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι καθόλου δίκαιη η συμφωνία όπως λέτε. Επίσης θα ήθελα τη γνώμη των νομικής υπηρεσίας. Το Μαρόκο έχει ποτέ ε, δηλώσει αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ε, χωρικά ύδατα της Δυτικής Σαχάρας και ανέπια είναι, είναι συμβατό με το διεθνές δίκαιο τα ευρωπαϊκά αλλιευτικά να δραστηριοποιηθούν εκεί. Ρωτώ λοιπόν, νομικά ποιος έχει δικαιώματα επί αυτής της ε, αποκλειστικής οικονομικής ε, ζώνης. Πέρα τα 200 ε, μίλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή φαίνεται ότι κρατάει πολύ ήδη. Και δεν θέλω να προσθέσω άλλα όσα ήδη υπόθηκαν, απλώ δύο στοιχεία. Το πραγματικό περιεχόμενο τη συμφωνία είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Ω προ αυτό, νομίζω ότι υπήρχαν εύλογε τάσει συμφωνία, διότι η αναλογία κόστου ωφελία και οι δυνατότητες μαζί με την χρηματική αντιπαροχή ήταν στοιχεία στα οποία υπήρξε συγκατάθεση. Ακόμη η ενδυνάμωση τη αρχή τη βιωσιμότητα που συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση ε, καλύπτεται καλύτερα και υπάρχει μετά και ένα δεύτερο ζήτημα. Η πολιτική ω προ τη Δυτική Σαχάρα. Εδώ δεν πιστεύω ότι κανείς στην αίθουσα σήμερα είναι περισσότερο ένθερμος υποστηρικτής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ότι εγώ ίδιο αναγνωρίζω ότι κάποιες φορές στο Κοινοβούλιο έχει σταθεί πάρα πολύ συζητώντα τα θέματα στην Επιτροπή Αλίας και όχι προωθώντα τα θέματα αυτά και στι υπόλοιπε επιτροπέ του Κοινοβουλίου. Στι διάφορε αρμόδιε επιτροπέ, όταν μιλούν για τη διεθνή μα πολιτική, τι εξωτερικέ μα υποθέσει, δεν αναλαμβάνονται πρωτοβουλίε για να μιλήσουμε για την περίπτωση και την πολιτική εξέλιξη τη Δυτική Σαχάρα. Ξέρουμε ότι πρόκειται για εδάφη τα οποία ε, τα διεκδικούν πάνω από 30 χρόνια και η Αλγερία και το Μαρόκο. Δεν λέω ότι αυτό το έδαφος θα πρέπει να θεωρείται ε, μαροκινό. Θα έπρεπε να δούμε όμως τι θα γίνεται με την ε, ε, τον αποκλεισμό ε, της Δυτικής Σαχάρας από τη Συμφωνία και το τι θα μπορούσαν να κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να επιληθεί το ζήτημα αυτό στο δυνατόν πιο σύντομα. Τώρα, η πορεία της αλίας σε αυτή την περιοχή είναι προφανώς ιδιαίτερα διδαλώδης εδώ οι αλληλευτικές δυνατότητες θα έπρεπε να δίνονται από τους, δυτικές, από τους διοικητές της Δυτικής Σαχάρας. Και στη συμφωνία το δεδομένο αυτό καλύπτεται από την αρχή της εδαφικής κατανομής. Εδαφική κατανομή των ωφελών της συμφωνίας. Τα οποία, την οποία μάλιστα εδαφική κατανομή θα την παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλει να την παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε, αν υπάρξει παραμικρή παραβίαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναστείλει τη συμφωνία. Μην ξεχνάμε και την άλλη όψη του νομίσματος, όσο καλή και αν θέλουμε να είμαστε. Να μην ξεχνάμε την τραγωδία στην οποία εξελίχθηκε η Αραβική Άνοιξη τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να ε, υλοποιηθούν πραγματικέ μεταρρυθμίσει στο Μαρόκο και στην Αλγερία. Μιλάμε για δύο καθεστώτα τη ε, Βόρεια Αφρική που είναι τα πλέον φιλοευρωπαϊκά τη περιοχή. Βρίσκονται στην πορεία του εκδημοκρατισμού του. και πρέπει σε αυτό να του ενισχύσουμε. Είναι πολύ σημαντικοί οι πολιτικοί εταίροι και συνεργάτε. Πρέπει να του αναγνωρίσουμε ω σημαντικού εμπορικού εταίρους. Έχουμε και άλλε συμφωνίε μαζί του. Έχουμε κυρώσει πρόσφατα γεωργικές συμφωνίε μαζί του. Ε, το ζήτημα της Σαχάρας είναι κάτι άλλο. Υπάρχουν οι Σαχαουοί και το πώς θα καθοριστεί βέβαια το πεπρωμένο του λαού αυτού είναι κάτι που θα πρέπει να το αναλάβουν στα χέρια τους οι ίδιοι οι έχουν λοιπόν όλα αυτά μια λογική, αλλά πρέπει να είμαστε και πραγματιστές. Θέλουμε να σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν έχουμε κάνει στο υπόλοιπο κοινοβούλιο αρκετές προσπάθειε για να έχει έναν ενεργό ρόλο στην επίλυση του, του ζητήματος της Δυτική Σαχάρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην βρίσκουμε τώρα το πρόσχημα με την αλληλευτική αυτή συμφωνία για να επιλύσουμε ένα τέτοιο ακαθόδε πολιτικό ζήτημα που παραμένει εδώ και χρόνια. Νομίζω λοιπόν ότι βελτιώσεις προφανώς μπορούν να επιφερθούν. Έχει γίνει ήδη ενδυνάμωση των ε, ανθρωπιστικών σκελών της συμφωνίας αυτής, αλλά νομίζω ότι η συμφωνία αυτή πρέπει να εγκριθεί. Και ήθελα πραγματικά να δώσω έμφαση και να τονίσω τόσο όσα υπόθηκαν, όσα υπόθηκαν σήμερα. Να θυμίσουμε ότι οι αλλιευτικοί πόροι που αλλιεύονται από τον Ευρωπαϊκό Στόλο στα ύδατα του Μαρόκου είναι λιγότερο από το 2% των συνολικών αποθεμάτων που αλλιεύονται στο Μαρόκο. Άρα οι πόροι αυτοί είναι βασικά αντικείμενο εκμετάλλευση του στόλου του Μαρόκου και άλλων στόλων από τον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να αναζητηθεί μια γρήγορη λύση για το πρόβλημα τη Δυτική Σαχάρα. Από αυτού που τα εκμεταλλεύονται περισσότερο. Ευχαριστώ κυρία Ρόντου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να πω κάτι θεμελιώδη στον κύριο Άγνιο. Κύριε Άγνιο, θα πρέπει τώρα να διαπιστώνετε ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι δειλό. Το Κοινοβούλιο κατάφερε να απορρίψει μια συμφωνία και να τη συζητάει εκ νέου. Εάν προσέξετε, θα δείτε ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν θα περάσει αυτή η νέα συμφωνία. Βλέπετε πόσες επικρίσεις διατυπώνονται. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβετε ότι πολλά ακόμη πρέπει να εξηγηθούν. Δεύτερη παρατήρηση προς εσάς. Όχι, σε εσάς απευθύνομαι. Να είστε σίγουροι ότι οι Βρετανοί φορολογούμενοι ε, και ε, τρώνε και ψάρια, δεν τρώνε μόνο κοτόπουλα για τη συμφωνία. Η απόρριψή μας είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλές θετικές αλλαγές στη νέα συμφωνία. Αλλά πιστεύω επίσης ότι πρέπει να συζητήσουμε ακόμη ορισμένα θέματα. Είμαι πεπισμένη ότι οι διατυπώσεις για τη Δυτική Σαχάρα δεν είναι επαρκώς συγκεκριμένες. Μιλάνε απλώς, ε, αναφέρει απλώς η συμφωνία για ε, την ανάγκη να είναι προς όφελος όλων των ε, πληθυσμών σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Δεν είναι επαρκής αυτή η διατύπωση. Η διατύπωση που είχαμε στην προηγούμενη συμφωνία πρέπει να βελτιωθεί. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς είναι δυνατόν να βελτιώσουμε, να κάνουμε πιο συγκεκριμένη αυτή τη διατύπωση. Να αναφέρεται για παράδειγμα, ότι θα πρέπει και ο πληθυσμό τη Δυτική Σαχάρα να ωφελείται από αυτή τη συμφωνία. Αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Κατά τα άλλα, ωστόσο, χαίρομαι για τις βελτιώσεις που ε, έχουν επέλθει. Ε, η ομάδα εργασίας μας ε, δεν έχει ασχοληθεί αναλυτικά ακόμη με τη συμφωνία αυτή και ξέρω ότι η περαιτέρω συζήτηση θα είναι ιδιαίτερα δυσχερή αν δεν επιληθούν όλα τα εκκρεμή θέματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρθία Ιέρρο. Ευχαριστώ κύριε Στίβενσον. Είναι δύσκολο να διαχωρίσουμε το λογικό από το συναισθηματικό. Δεν το λέω για όσους διαφορούν, διαφωνούν με μένα. Εγώ είμαι πάντα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το άλλο θέμα είναι πώς ορίζει το διεθνές δίκαιο την αυτοδιάθεση. Ξέρετε ότι εδώ υπάρχει μια διχογνωμία εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά δεν νομίζω ότι μια εμπορική συμφωνία για την αλληλεία είναι η καλύτερη δυνατότητα αντιμετώπισης του, θέματο, του θέματος αυτού. Δεν θα ήταν σκόπιμο και να καταψηφίσουμε για παράδειγμα τη συμφωνία με τη Μαυριτανία διότι και η Μαυριτανία ε, αλλιεύει σε ύδατα που είναι ε, έξω από κατεχόμενες περιοχές λέγοντας ότι είναι ιστορικό τους δικαίωμα. Και άλλες συμφωνίες έχουμε με άλλες χώρες που δεν σέβονται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν θέλουμε να είμαστε λογικοί, μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις, αλλά ειλικρινά είναι σαφής η κατάσταση. Ενάμιση χρόνο τώρα εργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές του Μαρόκου για να ε, λάβουν υπόψη το ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Ακούγοντας τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την εισηγήτριά μας και άλλους συναδέλφους η νέα συμφωνία βελτιώνει ουσιοδός την κατάσταση και για θέματα που μας αφορούν ιδιαίτερα ως Ευρώπη. Ξέρετε λοιπόν ότι ε, θα υπάρξουν μεγάλες βλάβες για όλους μας και για τα σκάφη μας. Και τα σκάφη μας προέρχονται από διάφορες χώρες, όχι μόνο από την Ισπανία. Εάν δεν μπορέσουμε να αλλιεύσουμε, και ξέρετε ότι έχει παραλύσει η οικονομία σε αυτές τις περιοχές. Ε, είμαστε σε τρομερή κρίση και μας ε, ζητιέται όλο και περισσότερη λιτότητα. Πρόκειται για μια συμφωνία στα πλαίσια πολύ πιο ευραίων σχέσεων που είναι αναγκαίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ έχω συνεργαστεί και εργαστεί πάντα για θέματα ασφάλειας και ανάπτυξης για τις σχέσεις μας με το Μαρόκο και νομίζω ότι οι συμφωνίες που έχουμε επιτύχει είναι επωφελείς για όλους μας και για την συνύπαρξη μεταξύ των δύο υπήρων και πλευρών. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν διότι στην αρχή ορισμένοι θεωρούσαν ότι ήταν υπερβολικές οι απαιτήσει του Μαρόκου έγινε διαπραγμάτευση και τώρα ε, η Ένωση θα πληρώσει 6 εκατομμύρια λιγότερο και απαιτείται περισσότερη συμμετοχή, οικονομική συμμετοχή από τους εφοπλιστές και υπάρχουν επίσης και ρήτρες διασφάλισης ούτως ώστε να ωφεληθεί και ο τοπικός πληθυσμός από τη νέα συμφωνία για να έχουν καλύτερη κατάρτιση, καλύτερη πρόσβαση στον κλάδο, καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Και καταλήγω με την αναφορά που έγινε από την Κομισιόν για την ε, ρήτρα που θα μας διασφαλίζει ότι θα παρακολουθούμε την εφαρμογή των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Αυτά μου αρκούν εμένα. Είναι καλή συμφωνία, πρέπει να τη στηρίξουμε. Τονίζω λοιπόν ότι ενώ ήμουν ιδιαίτερα αρνητική στο παρελθόν, τώρα όμως επειδή εδώ έχουμε μια εμπορική συμφωνία, δεν είμαστε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, Κοιτάξτε, αυτά είναι για αλλού. Και οι χώρες σας επίσης έχουν ευθύνη όταν έχουν, ε, για παράδειγμα, όταν συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, εκεί να τα πούν αυτά, όχι εδώ σε μια εμπορική συμφωνία για την Σας παρακαλώ, σέβομαι όλες τις απόψεις, αλλά και εγώ θέλω να γίνετε σεβαστή η δική μου και τονίζω Κοιτάξτε, σε πολλές άλλες περιπτώσεις που θα έπρεπε να έχουν τεθεί αυτά τα θέματα, εγώ δεν άκουσα να τίθενται. Το θέμα είναι περίπλοκο, πρέπει να καταλήξουμε. Όχι για αυτό το θέμα, αλλά και για πολλά άλλα, όχι μόνο για αυτό το θέμα. Δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή σε μια συμφωνία για την αλία. Δεν είναι δυνατόν να τίθεται τέτοια γενικότερα θέματα για να αποφεύγεται η υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας. Ευχαριστώ. Η κυρία Τόμας. Όχι, όχι, καλώς. Ο κύριος Τόρβαλτς. Ευχαριστώ όταν μιλάμε για το Μαρόκο. Ξαναλέμε τα ίδια. Άλλη μια φορά τα ίδια. Όποιος έχει δει την ταινία Κασαμπλάνκα ξέρει ότι η σωστή παράθεση δεν είναι play it again Sam αλλά play it Και περί τίνος πρόκειται, περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης θυμάμαι και μια όπερα του Μπιζέ, την όπερα Κάρμεντ. και η κυρία Φράγα λέγεται Κάρμεν. Δεν ξέρω τώρα εγώ θα είμαι ο Εσκαμίγιο ή ο Ντον Χωσέ. Θα δούμε τι ρόλο θα παίξω. Λοιπόν, θα είμαι σύντομος. Οι Ηνωμένε Πολιτείε όταν υπογράφουν ε, συμφωνίες Εξαιρούν πάντα την Δυτική Σαχάρα. Δεν υποστηρίζω πάντα τις ΗΠΑ, αλλά σε αυτό το θέμα νομίζω ότι έχουν δίκιο. Και αυτά που είπε η κυρία Λοβίν, ότι πρέπει να ζητήσουμε νομική γνωμοδότηση, νομίζω πως θα ήταν σκόπιμο να το κάνουμε αυτή τη στιγμή για αυτό το θέμα. Ενδιαφέρουσα επίσης η ερώτηση εάν ε, εποφελούμεθα αρκετά οικονομικά από αυτή τη συμφωνία. Μήπως αυτή η συμφωνία είναι επιδότηση για τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους και τους αλλιευτικούς τους στόλους. Μα θα έπρεπε να, έχουμε, να, να λάβουν κάποια ενίσχυση αυτές οι δύο χώρες. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε και τους Έλληνες ως Ευρωπαίοι είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες. Όχι ανοήτως να ε, εξετάζουμε μόνο εθνικά συμφέροντα. Δεν ήταν ε, προσωπικό, δεν έχετε προσωπικό για σας ε, φίλε μου, όχι, όχι, και στη Φιλανδία και για τη Φιλανδία θα μπορούσα να μιλήσω. Λοιπόν, είναι εδώ η Κάρμεν, θα δουλέψουμε μαζί θα τραγουδήσουμε μαζί αλλά πρέπει να ε, ε, προσέξουμε πολύ και τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σύντομα κύριε Καπούλας παρακαλώ. Παρακαλώ δεν θέλω να κάνουμε δεύτερο γύρο. Απλώς κάτι που υπόθηκε μόλις τώρα. Κανένα πορτογαλικό συμφέρον δεν αφορά αυτή τη συμφωνία. Ε, έχει 7 σκάφη στο Μαρόκο Πορτογαλία μόλις. Μιλάμε για πελαγική αλεία. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα συμφέρον από τη χώρα μου για την συμφωνία με το Μαρόκο. Ήθελα λοιπόν να το καταστήσω σαφές. Ε, me... Ωραία. Να πάρω και εγώ το λόγο. Ας θυμηθούμε ότι είμαστε Επιτροπή Αλίας, όπως είπε και ο κύριος Καπούλα Σάντος. Συζητήσαμε τα πάντα σήμερα το πρωί. Ανάπτυξη, ανθρώπινα δικαιώματα, δημόσιο διεθνές, πολυσάριο. Ο κύριος Τόρβαλτς μας μίλησε ακόμη και για όπερα και ταινίες του Humphrey Bogart. Μία πολύπλευρη λοιπόν συζήτηση και ωφέλιμη. Είμαστε Επιτροπή Αλίας ωστόσο. Αναβάλαμε, ε, αναστήλαμε αυτό το πρωτόκολλο σε μια προηγούμενη περίπτωση όπως ξέρετε αυτό κόστισε θέσεις εργασίας στους αλληλείς μας που αιώνες τώρα αλλιεύουν σε αυτή την περιοχή αλλά αυτό είχε ως συνέπεια την απώλεια θέσεων εργασίας και για το λαό της ε, Δυτικής Σαχάρας. Κύριε Άγνιου, ακούστε το εξής. Υπήρχε ένα σκοτσέζικο αλλιευτικό εκεί. Ήταν ένα από τα λίγα που με βάση το, την προηγούμενη συμφωνία εκφόρτωνε πελαϊκά είδη στην Τάκα και ο καπετάνιος έδινε έτσι δουλειά σε 300 γυναίκες της Δυτικής Σαχάρας, τις οποίες είχε καταρτήσει και με δικά του έξοδα είχε φτιάξει αυτή την επιχείρηση που απασχολούσε λοιπόν ε, εργαζόμενους από τη Δυτική Σαχάρα. Όλοι αυτοί που λένε ότι επειδή ψαρεύουμε σε ύδατα κατεχόμενης περιοχής δεν ε, βοηθάμε τον πληθυσμό της Δυτικής Σαχάρας, γιατί δεν ε, συζητήσαμε τον Πολυσάριο. Αυτοί ψήφισαν μέσω αυτής της στάσης τους ε, για ανεργία σε αυτή την περιοχή, στη Δυτική Σαχάρα. Έτσι προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουν δικαίωμα να εργάζονται οι άνθρωποι στη Δυτική Σαχάρα. Όπως είπε και η κυρία Πατράου. Όπως είπαν και άλλοι. 1% των αλλιευμάτων στα νερά του Μαρόκου της Δυτικής Σαχάρας αλλιεύονται από δικά μας σκάφη. Αλλά εάν εμείς δεν αλλιεύσουμε αυτό το 1%, και υποθέτω ότι εσείς θα καταψηφίσετε αυτή τη συμφωνία για άλλη μια φορά. Εάν εμείς λοιπόν δεν αλλιεύσουμε, αυτά τα αλλιεύματα θα τα δώσουν στους Κινέζους και τους Ρώσους που είναι ήδη παρόντες. Και επειδή υπάρχει ζήτηση στην Ευρώπη για αλλιείς, θα αγοράζουμε εμείς αυτά τα αλλιεύματα από τα βρώμικα, κινέζικα και ρώσικα αλλιευτικά και θα πληρώνουμε τους Ρώσους και τους Κινέζους. Και ξέρετε, αυτά τα σκάφη δεν δίνουν μία για τη Δυτική Σαχάρα, δεν εκφορτώνουν για κατεργασία και μεταποίηση καθόλου αλλιεύματα εκεί, δεν θα δώσουν καμία θέση εργασίας στους Σαχαράου και το λαό της δικής Σαχάρας, θα μεταφέρουν, θα μεταφορτώσουν εν πλώ τα αλλιεύματα αυτά. Αυτό θέλετε. Όχι, όχι, όλοι μιλήσανε και θα πρέπει να κλείσει η συζήτηση για να δώσω το λόγο στον κύριο Ντεπίπερ. Κύριε Στίβενσον, επειδή μου μιλήσατε απευθείας, δύο δευτερόλεπτα. Όχι, δεν απευθυνόμουν σε εσά προσωπικά. Μιλούσα για διάφορους συναδέλφους που ήταν τελείως αντίθετοι με το πρωτόκολλο. Όλοι έχουν δικαίωμα να δευτερολογήσουν, αλλά τώρα δεν μπορούμε να ξαναρχίσουμε από την αρχή τη συζήτηση. Όλοι είχαν δικαίωμα έκφραση. Ε, κοιτάξτε, θα ήθελα πάρα πολύ να τι δω αυτέ τι γυναίκε, αν μου είχαν επιτρέψει να κάνω την επίσκεψη, μου. Αλλά ήταν επίσημη απαγορεύση. Κοιτάξτε, έγινε ο σκύπερ αυτού του σκάφου, ο πλοηγός έκανε ταινία, γύρισε, τράβηξε βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε ευρέω. Τώρα αν δεν έτυχε να το δείτε εσεί, λυπούμε αλλά έδειχνε τις γυναίκες αυτές της Δυτικής Σαχάρας να δουλεύουν στην Τάκουα. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνεργοι ανέκαθεν. Αυτό το νέο πρωτόκολλο, αυτή η νέα εταιρική συμφωνία θα τους ξαναδώσει δουλειές. Και μπορούμε να εισάγουμε καθαρά εντό εισαγωγικών ψάρια που έχουν αλλιεύσει δικοί μας ψαράδες απασχολώντας ναυτιλωμένους από το Μαρόκο και τη Δυτική Σαχάρα θα τα εισάγουμε αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ένα πράγμα που θα ήθελα οπωσδήποτε να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχουν στοιχεία στη συμφωνία αυτή για την κατανομή των αλλιευμάτων. Από την ε, Σκοτία στέλνουμε πελαγικά σκάφη στην Δυτική Σαχάρα. Αλλά δεν θα το κάνουμε αν δεν παίρνουμε κάτι από τα αλλιεύματα. Ο πληγός μου είπε ότι δεν μπορεί, ο καπετάνιος μου ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ε, συγκεκριμένα στοιχεία. Ποιος θα πάρει τι και βάσει ποιων κριτηρίων. Βάσει του παλιού πρωτοκόλλου, τα Ολλανδικά σκάφη έπαιρναν το μεγαλύτερο μέρος των αλλιευμάτων. Και ήταν πολύ μεγάλος όγκος για να μπορέσουν να τα εκφορτώσουν στα τοπικά λιμάνια τα κρατούσαν στη θάλασσα. Τώρα ξέρω ότι τα λιμάνια έχουν βελτιωθεί, περισσότερα σκάφη θα μπορούν να εκφορτώνουν και αυτό είναι καλό βέβαια. Αλλά ενώ ήμουν αντίθετο με την αναστολή του προηγούμενου πρωτοκόλλου, έχοντα τώρα ακούσει τα όσα είπαν η Συγήτρια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι τόσο σημαντικέ βελτιώσει που έχουν επιφερθεί, νομίζω συνολικά άξιζε τον κόπο διότι εάν θέλουμε να ωφελήσουμε τους ανθρώπους της Δυτικής Σαχάρας και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας εκεί, σίγουρα πρέπει να υπάρξει τέτοια εταιρική σχέση. Και αυτή τη συμφωνία αξίζει να την στηρίξουμε. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο, κυρία Ρόντουστ και η κυρία Λέβιν. Μην ε, ξαναρχίσουμε όλη τη συζήτηση την αρχή. Ε, όχι, όχι, όχι, όχι, Στιούαρτ. Νομίζω ότι ε, για λόγους διαδικαστικούς πρέπει ε, ε, να λέτε πότε κλείνει ο κατάλογος ομιλητών. Είχα ζητήσει το λόγο πριν κλείσω ο κατάλογος ομιλητών. Κοιτάξτε. Ακούω ορισμένα πράγματα τα οποία, με τα οποία δεν συμφωνώ. Ως Επιτροπή Αιλίας φυσικά έχουμε δικαιώματα και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να προσέξουμε να εφαρμόζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και αν δεν εφαρμόζονται τότε πρέπει να σκεφτούμε με τα μέσα που έχουμε, τι δυνατότητε που έχουμε στη διάθεσή μα, τι μπορούμε να κάνουμε για να επιβάλλουμε την εφαρμογή του. Και μια τέτοια συμφωνία είναι ένα τέτοιο μέσο, μια τέτοια δυνατότητα. Και πρέπει να ε, σκεφτούμε τι θα την κάνουμε, αυτή τη συμφωνία. Θα πρέπει να σκεφτούμε. Μήπως θα μπορούσαμε να υπογράψουμε και συμφωνία αλλιές και με τη Συρία. Γιατί είναι εμπορική συμφωνία. Έχουμε ευθύνη και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας παρακαλώ, στη συζήτηση να τα σκέφτεστε αυτά τα πράγματα. Γιατί αλλιώ θέτουμε το ερώτημα είναι δημοκρατικός ο τρόπος ε, που επιχειρηματολογούμε. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Η συζήτηση σήμερα ε, ήταν οριακή από ορισμένες απόψεις σήμερα. Ευχαριστώ που ήσασταν σύντομοι. Η Ισοβέλ. Ή δυσκολίασα. Θα ήθελα να συναντώ με αυτές τις ε, γυναίκες και τους φίλους σας και όλους όσους επενδύουν στη Δυτική Σαχάρα αν θα μπορούσαμε να μπούμε σε αυτή την περιοχή. Και να θυμάστε επίση ότι προσπαθήσαμε ω επίσημα την προσωπία να πάμε στη Δική Σαχάρα και μα το αρνήθηκαν. Βέβαια, εδώ δεν πρέπει να συζητάμε πολιτική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί εδώ είναι η Επιτροπή Αλία. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, δεν είμαστε ειδικοί για θέματα αλία. Είμαστε πολιτικοί και τα πάντα είναι πολιτικοί. Τα τρόφιμα, ο αέρα που αναπνέουμε, το περιβάλλον είναι θέματα πολιτικής. Ο πρόεδρος. Ωραία, μετά από αυτήν την αναλυτική συμφωνία, ε, συζήτηση, κύριε Ντεπίπερ, ε, ίσως θα χρειαστείτε κάποιο χρόνο για να απαντήσετε. Λοιπόν, μου δώσετε αρκετά στοιχεία για να σας κάνω παρουσιάσεις και να συζητάμε μια ημέρα ολόκληρη. Θα αξιοποιήσω τις σημειώσεις μου και θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω λίγο αυτά που ακούστηκαν και να κωδικοποιήσω την απάντησή μου. Πρώτα απ' όλα να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο κ. Σάντο και εσεί κ. Στίβεν. Σε σχέση με το ερώτημα του κ. Άγνιου, θέλω να ε, διευκρινίσω μια παρεξήγηση. Εδώ δεν μιλάμε για τον στόλο της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Εδώ είναι μια συμφωνία από την οποία απευθολούνται βρετανικά σκάφη, ε, πολωνικά Ολλανδικά. Δεν έχω υπολογίσει επακριβώ, αλλά αν δείτε τις ποσότητες, ε, η κατανομή είναι πολύ πιο διαφοροποιημένη. Υπάρχουν πολλοί και διάφοροι στόλοι που θα υποφεληθούν. Και για να απαντήσω σε αυτό που είπατε κύριε Στίβενς για την κατανομή, αυτό είναι μια απόφαση του Συμβουλίου, την οποία θα διευκολύνουμε, θα προφροντίσουμε να βασίζεται στα διαφορετικές, στους διαφορετικούς τόλους. Και πράγματι, τα βρετανικά λιευτικά δραστηριοποιούνται έντονα στην περιοχή και θα υποφεληθούν από αυτό το πρωτόκολλο. Αυτό τεχνική απάντηση. Ετέθησαν κάποια πολλά εύστοχα ερωτήματα για τη γεωγραφική κατανομή και για την παρακολούθηση και για το αν θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τη διατύπωση. Το εξετάσαμε από όλες τις πιθανές σκοπιές το ερώτημα όμως νομίζω, το βασικό, είναι αν έχουμε πραγματικά τον έλεγχο και την εποπτεία της κατάστασης. Και υπάρχει μια ρήτρα που μας διευκολύνει να το έχουμε αυτό. Αυτή η ρήτρα θα μας ε, δώσει τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε μια διαδικασία και μετά σταδιακά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να λαμβάνουμε εκθέσεις ορθή γεωγραφική κατανομή είναι προαπαιτούμενο για να συνεχίζεται η εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Άρα η απάντησή μου είναι η εξή. Μπορούμε να αλλάξουμε τώρα τη διατύπωση, ε, θα έλεγα ότι μάλλον όχι. Έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών διαπραγματεύσεων. Αλλά μας ικανοποιεί αυτή η διατύπωση και μπορούμε να εμπιστευτούμε τη διαδικασία, μάλλον ναι θα έλεγα. στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε κάτι, να ξεκινήσει μια διαδικασία και αν στην πορεία δεν μας ικανοποιεί, πιθανώς να ε, τροποποιήσουμε τη στάση μας. Θα γίνεται λοιπόν προοδευτικά αυτή η εφαρμογή της συμφωνίας και θα εξελιχθεί στη διάρκεια του χρόνου η συνεργασία μας, θα μπορέσουμε έτσι να επιτύχουμε αυτό που θέλουμε. Τώρα για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενδιαφέρουσα συζήτηση. και συναισθηματική ορισμένες περιπτώσεις. Προφανώς είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Προφανώς και θέλουμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα ως κοινοβούλιο, εάν κρίνετε ότι υπάρχουν παραβιάσεις οι οποίες θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε αναστολή της συμφωνίας, ε, θέλουμε να το εξασφαλίσουμε αυτό. Αλλά δεν συμφωνώ καθόλου μαζί σας ότι αυτό είναι νεφελώδες και σαφές. Και θα σας εξηγήσω ακριβώς πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτή η διαδικασία αναστολής. να πω επίσης ότι άκουσα διάφορους να με προτρέπουν να λύσουμε το ζήτημα. Ε, μεγάλη τιμή μου περιποιείται, λες και θα μπορούσα να λύσω το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας και δεν το έκανα. Νομίζω αυτά τα πράγματα επιλύονται σε άλλο επίπεδο. Δεν υπονοώ ότι δεν πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τις προσπάθειες που γίνονται σε άλλα επίπεδα ή ε, να τα αξιοποιούμε και να τα λαμβάνουμε υπόψη μας όταν χαράσουμε πολιτικές, όπως για παράδειγμα αυτό το πρωτόκολλο, αλλά ε, νομίζω δεν είχα την εντολή να επιλύσω το εδαφικό πρόβλημα της περιοχής. Και αυτό μάλλον ξεπερνάει και τις ε, δυνατότητες μας. Οι αρμοδιότητες οι μας είναι η αλία. Δεν είμαστε ειδικοί σε θέματα ανθρωπινών δικαιωμάτων, απλώ δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε το Κοινοβούλιο, εσείς, να ε, αξιολογήσετε την κατάσταση και να ε, καταλήξετε σε συμπεράσματα. Τώρα, για το θέμα της αξιοποίηση των πορών και το ζήτημα της βιώσιμης αξιοποίησης τους, πρόκειται για πόρου οι οποίοι πρέπει να ανανεώνονται, το Εάν δεν πάμε εμεί το πλεόνασμα της αλίας θα το αλλιεύσουν άλλοι στόλοι. Το πλεόνασμα είναι ακριβώς εκείνη η ποσότητα ψαριών που μπορεί να αλλιευθεί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο σε καμία περίπτωση ε, η ισορροπία του περιβάλλοντος, η φυσική πόρη. Από πολλοί είπαν ή υπονόησαν ότι ε, αυτό το πρωτόκολλο πρέπει να περιοριστεί στα θέματα της αλίας και συμφωνώ πλήρως. Αλλά εάν διαπιστωθεί παραβίαση ανθρωπινών δικαιωμάτων, έχουμε τη δυνατότητα να αναστείλουμε την εφαρμογή του. Και να σας εξηγήσω λοιπόν τώρα τη διαδικασία. Επίσης δεν συμφωνώ με αυτό που είπατε ότι απλώς παραπέμπουμε σε μια άλλη συμφωνία. Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο το οποίο εξειδικεύει τη Γενική Συμφωνία Σύνδεσης. Λοιπόν, στο πρωτόκολλο Αλίας υπάρχει μία αναφορά στο βασικό κείμενο, στη Συμφωνία Σύνδεσης. Και αυτή η αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θεμελιώδης, είναι ουσιώδες στοιχείο της Συμφωνίας Σύνδεσης. Εξειδικεύουμε λοιπόν αυτό το ουσιώδες στοιχείο της Συμφωνίας Σύνδεσης. Τι λέμε, να αυτό το ουσιώδες στοιχείο της Συμφωνίας Σύνδεσης είναι επίσης ουσιώδες στοιχείο του πρωτοκόλου. Και στο άρθρο 8 του πρωτοκόλου προβλέπεται διαδικασία σε περίπτωση ε, διαφωνίας αναφερόμαστε ρητά στα ανθρώπινα δικαιώματα και λέγεται ότι σε περίπτωση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να ανασταλεί η εφαρμογή του πρωτοκόλου. Άρα δεν είναι καθόλου νεφελώδες, καθόλου ασαφές. Είναι ξεκάθαρο ότι σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των δημοκρατικών αρχών, εφόσον διαπιστωθεί αυτή η παραβίαση, μπορεί μέσω του άρθρου 8 και 1 να αναστελεί η εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δεν νομίζω χρειάζεται να μπω και σε άλλε λεπτομέρειες και απάντησα στα βασικά. Ευχαριστώ κυρία Φράγα. Είναι η τέταρτη ομιλία σας, Ιζαμπέλα. Θα το ξανασυζητήσουμε όταν η συγγήτρια θα υποβάλει την έκθεσή της. Γιατί κλείσαν το κατάλληλο των ομιλητών. Ε, έκανα δύο ερωτήσεις στην Επιτροπή. Μία. Πώς θα παρακολουθήσουν στο μέλλον τη συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και το δεύτερο, το Μαρόκο έχει διεκδικήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη επί των ε, υδάτων της ε, Δυτικής Σαχάρας. Η Επιτροπή όταν είπα ότι ελπίζουμε ε, να είμαστε ειδικοί για θέματα αλίας, δεν είμαστε ειδικοί για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν εμείς θα στείλουμε αποστολή να ε, ε, ελέγξει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σας παρακαλώ να περιμένετε να σας δώσω το λόγο. Η ερώτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, για την οικονομική ζώνη, αποκλειστική οικονομική ζώνη, είναι περίπλοκο θέμα που θεωρούσε ότι απευθύνεται στι νομικέ υπηρεσίε. Θα απευθυνθώ στι νομικέ υπηρεσίε. Ωραία, καλό να συμπεριληφθεί η γνωμοδότηση και των ε, νομικών υπηρεσιών. Ίσως θα μπορούσε ε, ο εκπρόσωπος νομικής υπηρεσίας. Ευχαριστώ σε αυτή τη φάση, σύμφωνα με τους ε, κανόνες, φυσικά με χαρά θα σας ε, δώσουμε ε, αιτιολογημένη απάντηση, αλλά δεν είμαι ε, σε αυτή τη φάση έτοιμος να σας δώσω τέτοια απάντηση τώρα. Ωραία. Να ζητήσουμε διευκρίνηση από τις νομικές υπηρεσίες να την έχουμε όταν θα υποβληθεί η έκθεση της συγγήτριας στην Επιτροπή. Πολύ σύντομα προς την Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έκανα δύο πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις στην Επιτροπή και δεν απαντήθηκε ούτε η μία ούτε η άλλη. Πρώτη, γιατί δεν εξαιρέθηκαν ε, τα ύδατα ε, κάτω από τον παράλληλο 1740. Είπε ότι θα μπορούσαμε να το επιλύσουμε ε, εξαιρώντας τα ύδατα που είναι κάτω από τον παράλληλο 2740. Πρόκειται για αλία. Εκεί είναι το όριο ε, κυριαρχίας του Μαρόκου με βάση το διεθνές δίκαιο. Γιατί να μην εξαιρέσουμε οτιδήποτε είναι κάτω από το 2740. Αυτό συμβαίνει με τις συμφωνίες μεταξύ, για παράδειγμα, Ηνωμένων Πολιτειών και Μαρόκου. Και η άλλη ερώτηση που δεν απαντήθηκε και την επαναλαμβάνω. Γιατί δεν ακούσατε τους νόμιμους εκπροσώπους του λαού Σαχαραουή είναι γνωστοί, συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις με τα Ηνωμένα Έθνη, είναι το μέτωπο Πολυσάριο. Γιατί δεν τους ε, συναντήσατε. Τώρα και άλλοι θέλουν το λόγο, αλλά έχει κλείσει ο κατάλογος. Δεν θα ξανακάνουμε ζήτηση για αυτό το θέμα πριν να έχουμε το σχέδιο έκθεση από την εισηγήτρια στην επόμενη συνάντησή μας. Αλλά ίσως θα μπορούσα να απαντήσω στο πρώτο τμήμα της ερώτησης του κ. Φερέιρα. Το προηγούμενο πρωτόκολλο που απορρίψαμε τόνισε ότι για τα πελαϊκά είδη τα μεγαλύτερα αποθέματα αυθονία ήταν στα ε, ύδατα της περιοχής Σαχαρουή ενώ τα αποθέματα στα ύδατα του Μαρόκου υφίστανται πίεση. Άρα μοιάζεται να λέτε γιατί απορρίπτουμε τη συμφωνία, γιατί δεν θέλουμε να αλλιεύσουμε εκεί που υπάρχει αυθονία και να συνεχίσουμε να αλλιεύουμε εκεί που δεν υπάρχει αυθονία. Νομίζω ότι είναι περίεργος τρόπος ε, να συμπεριφέρεται κανείς στην Επιτροπή Αλίας. Θα προτιμούσα να ασχολούμεθα κυρίω με ε, θέματα αλίας. Κύριε Ντεπίπερ, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Μα νομίζω ότι ήδη απαντήσατε κύριε Πρόεδρε. Αυτό που είπατε είναι ένα επιχείρημα γιατί δεν εξαιρέσαμε κάποια περιοχή. Η εντολή μας ήταν να ασχοληθούμε με όλα τα ύδατα. Γιατί δεν συναντήσαμε τους εκπροσώπους του λαού της Δυτικής Αχάρας. Βεβαίως τους είδαμε. Και μας εξέφρασαν σαφώς τις απόψεις τους. Πρόεδρος. Και τον τελευταίο λόγο η εισηγήτρια. Ευχαριστώ. εν μέρη τη συζήτηση αυτή την έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Αν θέλαμε να επιλύσουμε το πρόβλημα της ε, Δυτικής Σαχάρας μέσω μιας συμφωνίας αλληλείας, θα ήταν πολύ εύκολο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θα λύσουμε το πρόβλημα της Δυτικής Σαχάρας μέσω αυτής της συμφωνίας. Είτε υπάρξει αυτή η συμφωνία είτε την απορρίψουμε. Δεν μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα της Δυτικής Σαχάρας στα πλαίσια τα δικά μας. Το πρωτόκολλο αυτό όπως έχει καταλήξει μετά από τις διαπραγματεύσεις, ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες κατευθύντριες γραμμές της διαπραγματευτικής εντολής του Συμβουλίου. Και αυτά που έλεγε το, το... η έκθεση Χάγκλουν και αυτά που έλεγε και το ψήφισμα Χάγκλουν και από μένα και το δικό μου ψήφισμα που ενέκρινε η Ολομέλεια. Για αυτά λοιπόν υπερασπίζομαι. Δεύτερον, να απαντήσω στην κυρία Ρόντους για τον κλάδο. Στο άρθρο 6 του προηγούμενου πρωτοκόλλου, που είναι ταυτόσιμο με το 6 του νέου έχει μια αλλαγή ε, εστίασης. Όπως είπε η κοινωνική υπηρεσία αυτό που πρέπει να εγγυηθούμε είναι να είναι διαφανείς οι επενδύσεις που θα γίνουν σε αυτή την περιοχή της Σαχάρας Τέτοιε επενδύσεις γίνονται, αλλά δεν αναγνωρίζονταν προηγουμένω. Τώρα όμως θα αναγνωρίζονται. Θα πρέπει να μας εξηγήσουν τι επενδύσεις γίνονται σε όλε τις περιοχές. Λυπάμαι που δεν μπόρεσε να πάει στην Δυτική Σαχάρα η κυρία Λοβίν. Αλλά εγώ έχω πάει στον Τάκλα πρώτη φορά, πήγα πριν από 15 χρόνια και όποιος πάει τώρα θα διαπιστώσει ότι οι επενδύσεις που έγιναν για την λιευτική ανάπτυξη της περιοχής είναι τρομερές. Στο άρθρο 6 ε, αναφέρεται πώς πρέπει να μας παρουσιάζουν ε, το τι κάνουν. Τα έκαναν και προηγουμένως δεν τα ανέφεραν. Και για να απαντήσω στην ερώτησή σας για την κατανομή, η πρόταση κατανομής των δυνατοτήτων αλίευσης, όπως είπε και ο κύριος Δευθυντής, η βιομηχανική ε, πελαγική αλία δεν ε, κατανέμει τις δυνατότητες του. Η Ολλανδία θα έχει περισσότερα προβλήματα <clears throat> γιατί υπάρχει ένα ανώτατο όριο δυναμικού που θα <clears throat> είναι δύσκολο λόγω αυτού του ανωτάτου ορίου να αλλιεύσουν τα σκάφη της ε, Ολλανδίας. Αυτά που είπε ο κύριος Χάγκρον είναι εντάξει. <clears throat> Είμαι Ισπανίδα. Υπάρχουν δύο εθνότητες που αλλιεύουν. Ε, συγγνώμη, 12, 12. Δεν είναι μόνο οι Ισπανοί που αλλιεύουν σε αυτή την περιοχή. Υπάρχει επίσης η μικρή κλίμακα αλία, ε, η ισπανική, αλλά η βιομηχανική δεν είναι ισπανική. Εγώ ως εισηγήτρια θέλω να υπερασπιστώ όλους όσους πρέπει να υπερασπιστώ. Ε, τονίζω λοιπόν ότι 12 εθνότητες. Είναι πολλές χώρες. Η Ισπανία στη βιομηχανική αλία εκπροσωπείται σε πολύ μικρό βαθμό. <clears throat> Δεν έχω προσωπικό συμφέρον Με ενδιαφέρουν όλα τα θέματα αυτά, είτε ενδιαφέρουν την Ισπανία είτε όχι. Γιατί είμαι ε, βαθιά πεπισμένη Ευρω, Ευρωπαίστρια, θέλω να υπερασπιστώ όλους όσους αλλιεύουν σε αυτή την περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φράγα, η παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης θα γίνει στις 4 Νοεμβρίου και η ψηφοφορία ε, στην έκθεση, στην Επιτροπή μας. Ε, φυσικά δεν υπάρχουν τροπολογίες, θα πρέπει να ψηφίσουμε περί κατά. Θα γίνει στις 27-28 Νοεμβρίου η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Θα αποφασιστεί πότε θα γίνει κατόπιν. Ευχαριστώ πολύ. Ας περάσουμε στο επόμενο θέμα, το σημείο 9. Ελπίζω να μην υπάρχει τόση ε, διαφωνία για την εταιρική συμφωνία με τον Καμπόν. Θα μας την παρουσιάσει ο εισηγητής μας, ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να πω σε αυτή τη φάση. Με την επιφύλαξη μιας πλέον ε, λεπτομερούς εξέτασης κάποιων στοιχείων Υπάρχουν κάποιες ημερομονίες για να προχωρήσουμε και νομίζω ότι θα πάρει την πορεία του και το πρωτόκολλο αυτό. Απλώς να καταγράψουμε ότι το πρωτόκολλο αυτό σκοπό έχει να αντικαταστήσει το προηγούμενο πρωτόκολλο, το οποίο εξέπνευσε το Δεκέμβριο του 2011, το οποίο ίσχυσε για έξι χρόνια μεταξύ 2011 και 2013 αυτό που συνέβη θα μπορούσε να το εξηγήσει καλύτερη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά δεν υπήρξε πρωτόκολλο γιατί προέκυψαν κάποια προβλήματα κατά τις διαπραγματεύσεις τότε, τα οποία είχαν να κάνουν περισσότερο με την ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τις σχετικές πτυχές. Περιλαμβάνονται κατά κάποιο τρόπο στην αλία θέματα που δεν αφορούν άμεσα την αλία. Αυτά όμως δεν απαντώνται μόνο στη συγκεκριμένη συμφωνία και σε άλλες. Εδώ Τις διαπραγματεύσεις με το Γκαμπόν αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα, όμως το εμπόδιο αυτό ξεπεράστηκε. Η ρήτρα δεν έχει πλέον την προηγούμενη αμφισημία και την ευρύτητα στην ερμηνεία που επέτρεπε η προηγούμενη διατύπωση. Οι εκπρόσωποι της Γκαμπών εκεί είχαν εντοπίσει τα προβλήματα, κάποιες πολιτικές εξελίξεις που είχαν να κάνουν με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν πολύ ασαφής ε, η προηγούμενη μορφή της ρήτρα. Τώρα νομίζω ότι έχει αποσαφινιστεί αυτό, αλλά θα τα εξηγήσει καλύτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε σχέση με τις δυνατότητες και τα ποσά, οι δυνατότητες συμπεριλαμβάνουν 27 άδειες για θυναλιευτικά και 8 για θυναλιευτικά όχι για τα παραγαδιάρικα επιφανείας όπως ε, προβλεπόταν στο προηγούμενο πρωτόκολλο με 16 άδειες. Αυτή η αλλαγή των παραγαδιάρικων επιφανείας έχει να κάνει με αυτά που μειώθηκαν ε, με όσα ίσχυαν μάλλον από το προηγούμενο πρωτόκολλο κάτι που θα επιδεινωνόταν ε, από την εσωτερική νομοθεσία του Γκαμπών, η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα και δεν επιτρέπει την αλίευση καρχαριών στα εθνικά της χωρικά ύδατα. Ως προς την οικονομική διάσταση προβλέπεται αντιπαροχή για την περίοδο ισχύς της συμφωνίας, τριετία δηλαδή, 1.350.000 ευρώ, εκ των οποίων τα χιλιάδες αφορούν την πρόσβαση στις περιοχές αλίας, τα 450 ε, ετησίως, τα υπόλοιπα 450 ετησίως για, τον για την τομεακή στήριξη. Μιλάμε για σημαντική αύξηση των κονδυλίων της χρηματικής αντιπαροχής, κυρίως ως προς την πρόσβαση στις περιοχές αλίας. Να επισημάνω εδώ ότι υπάρχει καλύτερη κατανομή του, της προηγούμενης όπου το 60% των κονδυλίων αφορούσαν την υποστήριξη της βιωσιμότητας στην ε, εθνική πολιτική αλίας που είχε καθορίσει τον Καμπόν, ένα ποσοστό που τώρα χρησιμοποιείται για την τομεακή στήριξη. Και σε σχέση με το συνολικό ποσό της οικονομικής αντιπαροχής, ε, είναι μικρότερο σχετικά το ποσό, 450.000 ευρώ ΥΟΣ, ε, είναι μικρότερη αναλογία σε σχέση με το σύνολο του ποσού. Αλλά αυτό είναι το μόνο σημείο στο οποίο ήθελα να εντοπίσω την προσοχή σα. Ούτω ή άλλω θα δούμε αν θα προκύψει κάτι άλλο μέχρι τη στιγμή που θα ψηφίσουμε για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Φερέιρα. Η κυρία Παλμπόα. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερος που έχουμε αυτή τη συμφωνία που είναι αιτιολογημένο, αιτιολογημένη, ισορροπημένη θα επιτρέψει σε όλα αυτά τα σκάφη να αλλιεύουν και υπάρχει και η οικονομική αντιστάθμιση που συμπεριλαμβάνει δικαίωμα πρόσβαση και την ανάπτυξη της πολιτικής στον τομέα που δεν έχουμε σε άλλες συμφωνίες. Η αύξηση της οικονομικής ε, αντιστάθμισης αυξάνει, είναι 42% και μειώνονται η ε, όγκη. Το 20% των ε, αλλιέων πρέπει να είναι από τις χώρες ΑΚΕ με προτίμηση για τους ε, αλλιείς από την ε, ακτή ελεφαντοστού. Είναι καλό για την ακτή ελεφαντοστού αλλά είναι σημαντικό λοιπόν τα σκάφη μας να μπορούν να αλλιεύσουν θα αναπτύξουμε έτσι τις δυνατότητές τους και θα επιβάλλουν και τις απαιτήσει που έχουμε. Τα προβλήματα πρέπει να τα επιλύσουμε. Χαιρετώ, χαιρετίζω λοιπόν την συμφωνία αυτή. Και θέλω να ζητήσω και κάτι ακόμη σε αυτή τη συμφωνία και γενικότερα. Οι συμφωνίες αυτές πρέπει να ε, περιλαμβάνουν καλύτερη διαβούλευση με τον τομέα από την αρχική διατύπωση των προτάσεων της Κομισιόν μέχρι την τελική συμφωνία. Ο κλάδος ε, το διεκδικεί συνέχεια αυτό και πρέπει να το βελτιώσουμε να υπάρχει καλύτερη διακυβέρνηση αυτών των ε, συμφωνιών. Ευχαριστώ κυρία Λοβίν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή που μας παρουσίασε την ε, συμφωνία. Δεν είχα χρόνο να τη μελετήσω, καταλεπτός. Πολύ ενδιαφέρον βρίσκω το γεγονός ότι το άρθρο 7.1 λέει σαφώς ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση των Καμπών σημειώσουν ότι υπήρξε παραβίαση των θεμελιωδών και βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως ορίζονται από άρθρο 9 της Συμφωνίας Κοτονού μπορεί να ανασταλεί η Συμφωνία. Άρα σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει μια σαφής ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι να κρυβόμαστε πίσω από άλλες συμφωνίες. Τώρα για τους καρχαρίες, αναφέρατε τους καρχαρίες, δεν υπάρχει ποσόστοση για τους καρχαρίες ιδιαίτερος, όπως τη συμφωνία με τη Μαδαγασκάρη, κάτι που το θεωρώ εγώ θετική εξέλιξη σε εκείνη τη συμφωνία. Η ερώτησή μου λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τι θα γίνει με τα παραλίευματα καρχαριών. Είναι ένα μείζον ζήτημα στην αλλιεύση τόνου. Έχετε να σχολιάσετε κάτι. Ευχαριστούμε κυρία Φράγκα. Συγχαίρω την Κομισιόν που μετά από το μπλοκάρισμα που είχε υπάρξει επειδή το Καμπόν δεν ήθελε να υπάρχει αυτή η ρήτρα τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ρεσιμότητα τελικά έγινε εφικτό να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά. Αυτό δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει η Κομισιόν τα θέματα αυτά. Το Γκαμπόν είναι σημαντικό για τον ε, θύνα μας ε, στόλο. Είναι σημαντικό λοιπόν όσο δυνατόν περισσότερες συμφωνίες να έχουμε για τον τόνο με όσο δυνατόν περισσότερες χώρες για να εξοπλίσουμε όλο το δυναμικό μας. Σημαντική αύξηση λοιπόν Ε, το τέλος που ήταν 35 προηγουμένως ε, ευρώ κατά τόνο να πάει, ε, πήγε τώρα 55, τόν, 55 ευρώ ανά τόνο. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι αυξάνεται κατά πολύ η συμβολή των εφοπλιστών. Αυτό είναι καλή εξέλιξη και τη χαιρετίζω. Ευχαριστούμε κύριο Δεπίπερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω τα περισσότερα από τα θετικά στοιχεία καλύφθηκαν από τον εισηγητή και από τους διάφορους βουλευτές που πήραν το λόγο, να μην τα επαναλάβω. Όντως υπήρχε τέλμα για πολύ καιρό επειδή τα ανθρώπινα δικαιώματα και ρευσιμότητα ήταν ένα ζήτημα διαφωνίας. Τώρα να απαντήσω σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που τέθηκαν. Εάν ο τομέας Τη Αλία συμμετείχε στι όλε συζητήσει. Βεβαίω, βεβαίω προσπαθήσαμε να έχουμε τι συνεισφορέ του. Συζητήσαμε και μαζί του και στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν στενή η συνεργασία μα. Λόγω χάρη κάτι που δεν είχε γίνει στο παρελθόν ήταν ότι τώρα απαντήσαμε και σε συγκεκριμένε προτάσει του ελληνικού τομέα. Το ερώτημα για του καρχαρίε. Επειδή δεν έχουμε τράτες, δεν είναι θέμα οι καρχαρίες. Στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Τώρα για την τομεακή στήριξη και το ποσό που θα κατευθυνθεί εκεί. Αυξήθηκε το ποσό της τομεακής στήριξης, αλλά όχι μόνο για να διατεθούν περισσότερα κονδύλια, όπως στην ακτή του ελεφαντοστού και σε άλλους εταίρους, ενδεχόμενους εταίρους μας στη Δυτική Αφρική, πρέπει να προσθεθεί τεχνική στήριξη, τεχνική συνεργασία σε πολλές περιπτώσεις. Στο πρωτόκολλο εδώ μπορείτε να δείτε σημαντικές βελτιώσεις. Αυτές που μας επιτρέπουν να βοηθήσουμε έμπρακτα την χώρα να καταπολεμήσει την παράνομη αναρχική λαθρέα με αυξημένη ικανότητα να παρακολουθούνται τα σκάφη, οπότε και τα πρότυπα με το ηλεκτρονικό σύστημα επιβολής εκθέσεων να ε, καλύπτονται. Αυτά προσπαθούμε να τα ενσωματώνουμε σε όλες μας τις συμφωνίες και είναι ένα μεγάλο ποσοτικό άλμα ποιότητας για τις αλληλευτικές δυνατότητες των εταίρων μας. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες για κάποιες ε, τεχνικές πτυχές που καλό θα ήταν να λυθούν, αλλά πραγματικά επειδή ήταν σωστή και αποτί... ήταν καλή αποτίμηση, ελπίζω να τύχει μεγάλη στήριξη η συμφωνία και να προχωρήσει. Πρόεδρος, ευχαριστούμε την Επιτροπή. Μία, μία αμφιλεγόμενη αλληλευτική συμφωνία είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη. Ο κύριος Φερέρα θα υποβάλει το σχέδιο εκθεσής του στις 27-28 Οκτωβρίου, στη, ε, Νοεμβρίου μάλλον, στις 29 Ιανουαρίου θα εξεταστεί και το Φεβρουάριο του 2014 θα περάσει στην Ολομέλεια. Να περάσουμε στα διάφορα, να θυμίσω στα μέλη της Task Force, της ομάδας δράσης, ότι δύο μίνι bus, δύο μίνι λεωφορεία θα φύγουν στις 12.30 ακριβώς από την είσοδο στις 12.30 γιατί αρχίζει η συνάντηση στο Συμβούλιο στις 12.45. Κάτι άλλο στα διάφορα που θα ήθελε να αναφέρει κάποιος. Όχι. Περνάμε στο σημείο 11. Ενημέρωση για τις συστάσεις των συντονιστών από την πρωινή μας συνεδρίαση. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο να πω. Επόμενη συνεδρίαση τώρα στο σημείο 12, 14 Οκτωβρίου από τις 4 ως τις 6.30 στις Βρυξέλλες. Κυρία Λέβιν. Πρόεδρε, ο ίδιος είπατε ότι θα ήταν καλή ιδέα να ρωτήσουμε την νομική υπηρεσία τι θα γίνει με το EEZ. Θα γίνει αυτό. Ναι. Συμφωνήσαμε η νομική υπηρεσία να ετοιμάσει έκθεση ώστε να ακολουθήσει παράλληλα και την ε, έκθεση του εισηγητή και την πορεία της για την αποκλειστική οικονομική ζώνη του Μαρόκου. Ωραία. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Τελείωσε η πρωινή μας συνεδρίαση.